Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die heutige Sitzung, die Καλώς ήρθατε στη σημερινή συνεδρίασή μα. Είναι η τελευταία πριν από τι ερηνές διακοπέ. Το θέμα σήμερα είναι για την καταπολέμηση των απατών. Απευθύνω το θερμό καλώ ορίσατε και στι χώρε ε, των εθνικών ε, και στους ε, βουλευτές συγγνώμη, των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων με του οποίου συναντήκαμε χθε θα έχουμε αργότερα και την παρουσίαση του σχεδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Όλαφ και τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα με παρουσία του Επιτρόπου κ. Έτιγκερ, ο, στον οποίο δίνω αμέσως το λόγο. Καλημέρα κυρίε και κύριοι, καλημέρα κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, αξιότιμες κυρίε και κύριοι του Όλαφ, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε σήμερα να μπορούμε να σας παρουσιάσουμε την πρότασή μας για την τροποποίηση του κανονισμού που διέπει τις εργασίες του Όλαφ. Να πω πρώτα ότι είναι η τελευταία κοινοβουλευτική υποχρέωση ενώπιόν σας και θα μπορέσω να σας παρουσιάσω και τον κύριο Άιλετ, τον γενικό μας διευθυντή, ο οποίος ανέλαβε την εκτέλεση καθηκόντων διευθυντού, γενικού διευθυντού μάλλον, του Όλαφ, σε σύντομο χρονικό διάστημα μπόρεσε να αποδώσει τα μέγιστα ο κύριος Ήλετ και απέναντί σας και προς τα έξω για την ε, πρόθεση των θεμάτων και για αυτά που έχω να σας πω σήμερα, δηλαδή για την τροποποίηση του κανονισμού Όλαφ. Δεύτερο έχω να πω ότι το έγγραφο εργασίας το οποίο έχετε συντάξει εσείς ως εισηγήτρια κυρία Πρόεδρε, κατά τη γνώμη μου είναι ένα πραγματικό έργο το οποίο πηγαίνει σε βάθος δεν έρχεται αντίθετο με τη δική μας πρόταση. Πολλά από, σας, τα, πολλά από όσα ε, προτείνετε εσείς βρίσκουν απήχηση και στα δικά μας. Ίσως εκεί που έχουμε τη διαφορά είναι το επίπεδο φιλοδοξίας, ας πούμε, ή το τι μπορεί να μείνει κανείς από το Συμβούλιο Υπουργό να το πω διαφορετικά. Θα χρησιμοποιήσω την ευκαιρία τη επίσκεψή μου μετά στο Συμβούλιο Υπουργών για να παρακαλέσω την Αυστριακή Προεδρία και να την προτρέψω να λάβει υπόψη τη την πρόταση που κάνουμε για την τροποποίηση του κανονισμού ω ένα από τα κέντρα βάρου. Διότι έχω βεβαίω κάθε κατανόηση και σεβασμό για την προσπάθεια προστασία των εξωτερικών συνόρων, αλλά και τούτο εδώ το θέμα είναι σημαντικό. Για μα έχει σημασία με το σχέδιο κανονισμού μας να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν μακρύτερα μέχρι τις ευρωεκλογέ, μέχρι δηλαδή το, την λήξη των κοινοβουλευτικών σας δραστηριοτήτων ή δυνατόν μάλιστα να καταλήξουμε και σε απόφαση, τουλάχιστον να γίνει μια πρώτη ανάγνωση. Διότι όλοι οι συμμετέχοντες και ιδίως ό,τι αφορά την οριοθέτηση των καθηκόντων του ΟΛΑΦ χρειάζονται ασφάλεια δικαίου και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αλλά και για την ανάπτυξη Ενό ισχυρού μηχανισμού, μια ισχυρή ομάδα του Όλαφ που να έχει ξεκάθαρα οριοθετημένα καθήκοντα και να υπάρχουν ξεκάθαρα, ε, ε, ξεκάθαρα ορισμένα καθήκοντα και των δύο αυτών φορέων, Όλαφ και η ΠΠΟ, δηλαδή Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αρχίσαμε με την Επιτροπή Προπολογισμών του Ευρωκοινοβουλίου, να συζητούμε δηλαδή το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο για την επόμενη δεκαετία και βλέπω και εδώ στενή διασύνδεση, διότι το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο θα είναι αξιόπιστο εάν εξασφαλίσει την συνέχιση παλαιών προγραμμάτων, την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων, θα είναι τότε αξιόπιστο μόνο όταν ο έλεγχος του προϋπολογισμού και η καταπολέμηση καταχρήσεων των ευρωπαϊκών κονδυλίων αντιμετωπίζονται από έναν αποδοτικό οργανισμό, Όλαφ, και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που θα διαθέτουν τις αναγκαίες αρμοδιότητες και εργαλεία. Γι' αυτό, άλλωστε, η μεταρρύθμιση του κανονισμού Όλαφ αποτελεί και μια συμβολή για έναν ισχυρό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για την επόμενη δεκαετία. Το 2017 συντάχθηκε η οδηγία για την ποινική δίωξη απατών. Η οδηγία PIF, PIF, καθώς και ο κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Άρα δύο σημαντικά θεμέλια. Η πρότασή μας σήμερα για την τροποποίηση του κανονισμού Όλαφ λαμβάνει υπόψη τις δύο αυτές σημαντικές εξελίξεις και τις συμπληρώνει. Θέλουμε δηλαδή να εξυγχρονίσουμε το πλαίσιο δραστηριοτήτων του Όλαφ και αυτό θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό. Γιατί χρειαζόμαστε γρήγορα το πλαίσιο επεξεργασία του κανονισμού ΟΛΑΒ. Λέω γρήγορα, διότι θέλω να καταδείξω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΟΛΑΦ αντιλαμβάνονται ότι η πρότασή μα δεν είναι ευέλτιστη. Δεν γίνονται δηλαδή τέλεια τα πράγματα με την πρότασή μα. Καθίσαμε και σκεφτήκαμε σοβαρά μαζί με τον τα ε, χρέη Γενικού Διευθυντού κ. Άιλετ, καθώς και με τον προκάτοχό του, πάρα πολλές ώρες. Και καταλήξαμε σε μια διαδικασία δύο φάσεων. Τώρα μια μικρή αναθεώρηση, η οποία θα εξυπηρετήσει κυρίως τον στόχο να διορθώσει όσα τεχνικά είναι δυνατόν, επειδή η ΕΠΟ βρίσκεται τώρα στη φάση της γένεσής της, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, Σα διαβεβαιώ όμως ότι στην επόμενη εντολή της, η ε, επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή, αμελητή και βασισμένη στο δικό σα έγγραφο εργασία θα προχωρήσει σε μεγαλύτερη τροποποίηση η οποία θα μπορέσει να γίνει χωρίς πλέον πίεση χρόνου να συζητηθεί και να ολοκληρωθεί 2020-2021. Δηλαδή τώρα προβάλλουμε την ταχεία λύση για την προσαρμογή στις ανάγκες και η μεγάλη λύση θα έλθει σε δύο θα έρθει αργότερα και θα είναι αυτές οι δύο φάσεις της συνολικής αναθεώρησης. Τώρα, η ταχεία λύση. Πρώτα, πρέπει να προσαρμόσουμε τις δραστηριότητες της Όλαφ στην ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, με τρόπο ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις και ασάφειες ό,τι αφορά την οριοθέτηση των λειτουργικών καθηκόντων τους. Εδώ χρειάζεται βιασύνη, χρειάζεται ταχύτητα, διότι ο κανονισμός Όλαφ δεν θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ πριν να ολοκληρωθεί και να αναλάβει δράσεις η Ευρωπαϊκή Αγγελία. Χρειαζόμαστε επίσης την ανανέωση αυτή του κανονισμού για να είναι ισχυρός, ισχυρό το αυτό το γραφείο δηλαδή καταπολέμησης άπατων να έχει διαφορετική εντολή από αυτό την, των, ε, της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και αυτά να αλληλοσυμπληρώνονται. Γι' αυτό και το νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να ξεκινά από την αξιολόγηση που έχουμε διεξαγάγει και στην βάση ε, εγγράφου και να βελτιωθεί. Οι προτινόμενες αλλαγές καταδεικνύουν την βούληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταθέσει πρόταση η οποία να μπορέσει να ολοκληρωθεί πριν να αναλάβει τα καθήκοντά τη Ευρωπαϊκή Αγγελία. Τώρα, η πρόταση έχει δύο σκέλη. Αφενό, η συνεργασία Όλαφ ή ΠΠΟ, από την άλλη μεριά, η αύξηση τη αποτελεσματικότητα των ερευνών του Όλαφ συνολικά. Όλαφ ή ΠΠΟ. Εμεί θεωρούμε την ίδρυση τη Ευρωπαϊκή Αγγελία θεμελιώδη ε, πρόοδο στην καταπολέμηση της απάτης στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Βεβαίως, η αυξηση τη αποτελεσματικοτητα των ερευνων του ολαφ συνολικα ολαφ η ππο εμει θεωρουμε την ιδρυση τη ευρωπαικη αγγελια θεμελιωδη προοδο στην καταπολεμηση τη απατηση στο ευρωπαικο επιπεδο βεβαιω η ιδρυση τη ευρωπαικη αγγελια δεν επιτρέπεται με κανένα τρόπο να μειώσει τις δραστηριότητες του Όλαφ. Δεν επιτρέπεται δηλαδή να οδηγήσει σε αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά τη επιχειρησιακή δράση του Όλαφ. Ο Όλαφ πρέπει να παραμείνει ισχυρός και λειτουργικός. Τη δυνατότητα ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να συμπληρώνουν οι έρευνε του Όλαφ. Όλαφ σε όλε τι χώρε θα διατηρήσει την εντολή του για την διερεύνηση διοικητικών υποθέσεων, εκτός δηλαδή των ποινικών, όπου υπάρχουν παρατυπίες που δεν αποτελούν απάτη. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι αρμοδία για διοικητικές παρατυπίες. Για να δώσω ένα παράδειγμα. Το 2016 93% περίπου όλων των καταγγελιών αναφέρονταν σε παρατυπίες που δεν αποτελούσαν απάτη, άρα δεν ήταν ποινικού χαρακτήρα. με συνολικό όγκο περίπου 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεύτερον, ο Όλαφ θα διεξάγει τις έρευνές του στις χώρες εκείνες μέλη που δεν συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό θα συνεχίσει απαράλλακτο, χωρίς απολύτως καμία μείωση. Τρίτο, στις περιπτώσεις ποινικά διοκόμενης απάτης. Στις χώρες εκείνες μέλη που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εκεί η Εισαγγελία και όλα θα συνεργάζονται. Οι μεν θα ενισχύουν τους δε στις προσπάθειές τους και αυτά στα πλαίσια των εντολών του κάθε οργανισμού. Για να συγχρονιστεί η νομική βάση του Όλαφ, η πρότασή μας προβλέπει νέες διατάξεις για σημαντικούς τομείς κλειδιά. Έχουμε περιλάβει διατάξεις που αναφέρονται στην ανταλλαγή πληροφοριών και τα ανάγουμε αυτά σε κεντρικό σημείο συνεργασίας Όλαφ και ΕΠΠΟ. Όλαφ και ΕΠΠΟ θα ανταλλάσσουν αμοιβαία πληροφορίες, θα πρέπει να συνεργάζονται σε πολλές περιπτώσεις ώστε να καθορίζουν ποια είναι η καλύτερη προσέγγιση που μπορεί να είναι ποινική, μπορεί να είναι διοικητικού χαρακτήρα ή μπορεί να έχει και τις δύο ιδιότητες. Εδώ βασιζόμαστε και στην καλή βούληση των επικεφαλής των δύο αυτών φορέων. Θα πρέπει να δείξουν δηλαδή, ιδίω στα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους, πόσο συνεργάσιμοι είναι και πόσο μπορεί αυτή η συνεργασία να είναι συνεκτική. Ένα κέριο σημείο θα είναι και το καθήκον του Όλαφ να θέτει υπόψη της εισαγγελία αμελητή στοιχεία, δεδομένα, στη βάση των οποίων μπορεί να ξεκινήσει μια ποινική δίωξη. Ο Όλαφ θα πρέπει, αυτή είναι η απόλυτη πεποίθησή μου, να γίνει κύρια πηγή πληροφοριών για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στην πρότασή μας Νομίζομαι ότι έχουμε επιτύχει μία ισορροπία ανάμεσα στο καθήκον άμεσης κοινοποίησης ενημέρωσης και της αναγκαιότητας σε ορισμένες περιπτώσεις ο Όλαφ να επαληθεύει πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει, να τις διασταυρώνει. Θα πρέπει λοιπόν, λέω το δυνατόν συντομότερο, να τίθεται υπόψη τη εισαγγελία ή πληροφορίε. Οι πληροφορίε αυτέ θα πρέπει να έχουν όμω μια επαρκή ποιότητα και να μην βασίζονται απλώ σε φήμε. Για να επικαλυφθεί η επικάλυψη εργασία και να υπάρξει η μέγιστη συμπληρωματικότητα με τι δραστηριότητε τη Ευρωπαϊκή Αγγελία, η μεταρρύθμιση μα προβλέπει διατάξει για την λειτουργικότητα του Όλαφ και για τις ε, διώξεις που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στις χώρες μέλη που συμμετέχουν θα πρέπει οι διοικητικές έρευνες του Όλαφ να επιτρέπουν την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων και την αποτροπή μεγαλύτερη ζημία για τα οικονομικά συμφέροντα τη Ένωση. Περιλαμβάνουμε και διατάξει για την αποφυγή επικαλύψεων και για τη συμπλήρωση των δραστηριοτήτων όπου αυτό είναι αναγκαίο. Εάν δηλαδή η διοικητική ανάκτηση πρέπει να γίνει άμεσα. Εάν υπάρχει, για παράδειγμα, κίνδυνος παραγραφής. Η, ε, η, τα διακινδυνευόμενα ποσά είναι πάρα πολύ υψηλά. Τροποποιήσεις επίσης που αναφέρονται στην εισαγγελία αναφέρονται στην υποστήριξη από πλευράς Όλαφ προς την εισαγγελία μετά από δική της αίτηση. Εάν δηλαδή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πάει και χτυπήσει την πόρτα του Όλαφ και ζητήσει αρρωγή έχουμε διατυπώσει τις διατάξεις του κανονισμού ή e PPO με τέτοιο τρόπο που απηχούνται ακριβώς. Η διατύπωση δηλαδή που βλέπετε στον κανονισμό ή e PPO βρίσκεται στο, και στον κανονισμό για τον Όλαφ. Θα έχει τη δυνατότητα λοιπόν ο Όλαφ να στηρίζει το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και με αντικειμενικές αναλύσεις και άλλες ε, παροχές δεδομένων. Η κυρία Πρόεδρος έχει τονίσει τη διαφορά μεταξύ των εντολών των δύο οργανισμών και τονίζει επίσης ότι οι δύο οργανισμοί θα πρέπει να εργάζονται συμπληρωματικά. Αυτό όμως σημαίνει ξεκάθαρη οριοθέτηση. Πέραν τώρα τη συνεργασία η ΠΠΟ Όλαφ. Ο Όλαφ θα συνεχίσει να διαθέτει ιδίαν εντολή και την οποία θα πρέπει να εκπληρεί. Και η πρότασή μας αναφέρεται και στοχεύει στην εξασφάλιση του ότι αυτό θα γίνει με, τον δυνατότερο αποτελεσματικό, με τον αποτελεσματικότερο μάλλον δυνατό τρόπο. Δεν προχωρούμε διότι θα ήταν πρόημο σε πλήρη αναδιάθρωση του κανονισμού του Όλαφ. Διότι αυτό δεν θα εξυπηρετούσε τον στόχο. Γνωρίζω ότι από εσά αξιότιμες κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές ότι εσείς προτιμάτε μια σε βάθος αναδιάρθρωση. Έχει εντοπίσει και άλλους τομείς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου αλλαγές θα ήταν σωστό να γίνουν. Όμως τώρα μάλλον να γίνει αυτό τώρα θα ήταν μάλλον υπερβολικά φιλόδοξο και γι' αυτό προτιμούμε αυτή την προσέγγιση σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση περιοριζόμαστε σε ορισμένες σημαντικές αλλά περιορισμένες αλλαγές που αναφέρονται στις έρευνες του Όλαφ και αυξάνουν την αποτελεσματικότητα των ερευνών αυτών. Η συνοχή των δραστηριοτήτων του Όλαφ στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παίζει και εδώ έναν σημαντικό ρόλο. Δεν μπορούμε δηλαδή να επιτρέψουμε στη, σε έναν οργανισμό, ευρωπαϊκό οργανισμό, το οποίο λειτουργία βασίζεται σε κανονισμό, να μπορεί να ασκεί τι δραστηριότητε του στι διάφορε χώρε μέλη με υποτελείω διαφορετικέ συνθήκε. Αυτή η απόκληση των συνθήκων στι διάφορε χώρε μέλη, μας απασχολεί και θέλουμε να την εναρμονίσουμε ή δυνατόν στην πρώτη αυτή φάση. Αναφέρομαι στις τροποποιήσεις ιδίως για τους επιτόπιους ελέγχους που αποτελούν και το σημαντικότερο μέσο που διαθέτει ο Όλαφ. Η πρότασή μας λέγει ότι γίνονται με εναρμονισμένο ομοιόμορφο τρόπο οι έρευνες του Όλαφ σε όλες τις χώρες μέλη. και προβλέπουμε και την υποστήριξη που δίνουν οι συντονιστικές αρχές των χωρών μελών στον Όλαφ. Από πλευρά λοιπόν αρχών, κρατικών αρχών, αρχών δηλαδή εθνικών ή και περιφερειακών. Στην πρότασή μας διευκρινίζεται και η εργαλειοθήκη που διαθέτει ο Όλαφ στην καταπολέμηση απατών ε, του φόρου κύκλου εργασιών. Και αυτό το έχετε τονίσει κυρία Γκρέσλε, στο έγγραφο εργασία σα. Επιθυμώ να τοποθετηθώ τώρα σύντομα για ορισμένε άλλε τροποποίησει. Στο έγγραφο εργασία της κυρίας Γκρέσλε προτείνεται περαιτέρω τροποποίηση στις διαδικαστικές εγγύησει αντιλαμβάνομαι το Κοινοβούλιο προσμετρά σημαντική σημασία, μεγάλη σημασία για ε, τούτο εδώ. Θα τα επεξεργαστούμε για να ενισχύσουμε τις διαδικαστικές εγγύσεις. Από την άλλη μεριά χρειαζόμαστε, σύμφωνα με την, με την άποψή μας τώρα, δεν χρειαζόμαστε μάλλον σε βάθος τροποποίηση στον κανονισμό 883 του 2013 θεσπίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα και με τον θεμελιώδη χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διοικητικού χαρακτήρα έρευνες γίνονται από τον Όλαφ στην βάση του διοικητικού δικαίου και όχι του ποινικού. Ο κατακαιρματισμός όμως του νομικού πλαισίου είναι σημαντικός. με, το, με τη συγχώνευση σε ένα νομοθέτημα του κανονισμού 883 καθώς και των υπολείπων ε, συναρμόδιων νομοθετημάτων. Γιατί υπάρχουν προβλήματα συνοχής ανάμεσα στις διάφορες νομικές βάσεις που διέπουν τι δραστηριότητε του Όλαφ και που έχουν αναπτυχθεί ιστορικά. Στη δεύτερη φάση λοιπόν θεωρούμε ότι αυτή η εναρμόνιση πρέπει να αποτελέσει το κύριο μέλημά μας πλήρης ενοποίηση των νομοθετημάτων που θεωρώ ότι είναι σημαντική, δεν μπορεί να επιτευχθεί κατά πάσα πιθανότητα μέχρι τον Μάιο του επομένου έτους, που είναι το χρονικό περιθώριο που διαθέτουμε. Και γι' αυτό θα είναι το δεύτερο σκαλί, η δεύτερη φάση στην διαδικασία αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε και άλλες περιπτώσεις, που έχουν και άλλες διατάξεις που χρειάζονται βελτίωση. Εμείς προτείνουμε ωστόσο μια ρεαλιστική προσέγγιση και αυτό κατά τη γνώμη μου συμβαδίζει με τις δικές σας προσδοκίες. Ολοκληρώνοντας, ο Όλαφ θα πρέπει να είναι στενός και αξιόπιστος συνεργάτης της ε, Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Ισότιμος εταίρος δηλαδή. Γι' αυτό το λόγο απαιτούνται ξεκάθαροι όροι συνεργασίας των δύο φορέων και μάλιστα να υπάρχουν πριν αρχίσει την άσκηση του έργου της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Γι' αυτό επισημαίνω και πάλι το επίγον, τον επίγοντα χαρακτήρα δηλαδή των διαδικασιών ενώπιον του σεβαστού σας ε, οργάνου, καθώς τα ίδια θα πω και στο Συμβούλιο των Υπουργών. Βασίζομαι στην δική σας συνεργασία και για την ε, προσπάθεια που θα κάνουμε μετά το 2020 για να συνεργαζόνται τα δύο αυτά όργανα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, λέει η Πρόεδρος, για την παρουσίαση της ε, νομικής βάσεως. Κύριε Επίτροπε, μιλήσατε για κοινά σημεία και για ενδεχόμενα ε, ενδεχόμενες δυσκολίες. Καλωσορίζω και τον κύριο Άιλετ, που είναι ο εκτελών καθήκοντα Γενικού Διευθυντού χαίρομαι για τους επένους. Παρούσα είναι και η Επιτροπή Εποπτείας του έργου του Όλαφ. Είμαι η συγγήτρια, θα σας απαντήσω κύριε Επίτροπε σε ορισμένα σημεία. Θεωρώ ότι έχουμε την ευκαιρία τώρα να ξεκαθαρίσουμε τις εντολές και της ΕΠΟ, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και του Όλαφ. Η εντολή του Όλαφ είναι οι διοικητικές έρευνες. Δεν είναι δυνατόν πλέον ο Όλαφ να προσπαθεί να αντιμετωπίζει ενδεχόμενες ποινικέ υποθέσεις απλώς με την εργαλειοθήκη των διοικητικών ερευνών. Προκύπτουν πολλά προβλήματα, ξεκινώντας από τα διαδικαστικά δικαιώματα των συμμετεχόντων μέχρι την έρευνα την οποία βεβαίως οφείλει να διεξαγάγει η εισαγγελία. Θεωρώ λοιπόν ότι οι επικαλύψεις αυτές, μάλλον οι συγκρούσεις αυτές αρμοδιοτήτων, καθώς και οι επικαλύψεις ενδεχομένως αργότερα πρέπει να αποφευθούν. Αυτό δεν είναι απλό. Πρέπει να αποφύγουμε και ενδεχόμενες μακροχρόνιες συγκρούσεις αρμοδιοτήτων μεταξύ Όλαφ και Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Πρέπει να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε την επιτυχία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, διότι θα είναι το πρώτο, το πρώτο όργανο στο επίπεδο της Ένωσης, το οποίο αφενός θα μπορεί να επιλέγει τις υποθέσεις με τις οποίες θα ασχολείται, αφετέρου δεν θα χρειάζεται δηλαδή να του τις ε, διαβιβάσει κανείς, και από την άλλη μεριά έχει και τα εργαλεία να δράσει. Δεν επιτρέπεται να δημιουργήσουμε δηλαδή άλλα όργανα τα οποία να αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες αυτές που δεν θα μπορεί να λάβει η ΕΠΟ. Ευχαρίστω λοιπόν να ασχοληθώ και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όταν θα υπάρξει και να φροντίσουμε να λειτουργήσει με τον τρόπο που πρέπει. Δηλαδή αυτό το πρόβλημα της ενδεχόμενης, καταστρα... της ενδεχόμενης ε, αποφυγής κάποιων ε, μπλοκαρισμάτων είναι απαραίτητο. Εφόσον δηλαδή αποφασίσει να ανοίξει μια υπόθεση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο Όλαφ θα πρέπει να μπορεί να διεξάγει έρευνα και μετά από αίτηση τη ε, ΕΠΟ, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εδώ δεν αρκεί η πρόταση τη Κομισιόν και θα χρειαστεί βελτίωση. Επίση υπάρχει δεκαήμερη προθεσμία μετά από ε, αίτημα του Όλαφ για να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό θα λειτουργήσει δύσκολα και δεν είμαι βεβαία ότι δεν πρέπει να κάνουμε εκεί κάποια βελτίωση. Και θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε ένα αυτόματο μηχανισμό ελέγχων για τη διεξαγωγή συμπληρωματικών ερευνών. Έχουμε και μία προθεσμία 30 ημερών προβολής ενστάσεως από την ΕΠΠΟ για την ανάληψη δράσεως από τον Όλαφ εδώ όμως παίζει ένα ρόλο η ΕΠΠΟ που κανονικά δεν τη ανήκει κατά τη γνώμη μας. Γιατί καλείται να αιτιολογήσει την ένσταση. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να κινείται αντίθετα η διαδικασία, δηλαδή ο Όλαφ να ζητεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να του επιτρέψει να διεξαγάγει την διοικητική έρευνα. Και να διαγραφεί η τριακονθήμερη προθεσμία. Υπάρχει και μια πρόταση για την πρόσβαση σε δεδομένα τραπεζικών λογαριασμών. Νομίζω ότι αυτή είναι υπερβολική, θα την εξετάσουμε προσεκτικά. Θα ζητήσουμε και τη γνώμη νομομαθών. Να δούμε τι θα μας πούν. Για τις διοικητικές έρευνες και τη διασύνδεση δηλαδή με τις δυνατότητες διεξαγωγή διοικητικών ερευνών στις χώρες μέλη, αυτό πρέπει να είναι διαβιέστατο. Επομένως θα χρειαστεί και βελτίωση της πρόσβασης πληροφοριών, της πρόσβασης πληροφορίες που διαθέτουν οι χώρες μέλη. Υπάρχουν ασθενή σημεία στον ε, παρόντα κανονισμό και μετά από την τελευταία αναθεώρηση του Όλαφ είχαν συζητηθεί αυτά. Σε αυτόν τον σύντομο κανονισμό Όλαφ δεν ξέρω αν θα προχωρήσουμε γρήγορα ή αργά. Θα προχωρήσουμε αργά γιατί και το Συμβούλιο Υπουργών κινείται αργά και δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τα πράγματα που συμβαίνουν εδώ στις Βρυξέλλες. Και ενδιαφέρονται οι υπουργοί μονάχα, τόσο, για, μονάχα για τόσα συμβαίνουν στις ε, μέλη. Θα ακούσουμε την κριτική και της ε, Εποπτικής Επιτροπής για την εκλογή της Review Unit στην ε, έκθεση. Εδώ νομίζω πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι πληροφορίε πρέπει να διαβιβάζονται αμελητή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μόλις ε, διαγνωστεί ενδεχόμενος ποινικό χαρακτήρας. Τα βασικά σημεία του κανονισμού ΕΠΟ μπορούν να αποτελέσουν κάποιο πρόβλημα όπως έγινε και ε, με την ΠΙΦ. Ε, και εννοώ εδώ τις τιμές, κατόφλια δηλαδή, τις κατώτερες τιμές τις κατώτατα ποσά, τα κατώτατα διακυβευόμενα ποσά δηλαδή. Και τι θα κάνουμε με όλες τις ποινικέ υποθέσεις που είναι κάτω των κατοφλίων των διακυβευόμενων ποσών. Έχουμε και άλλες ασαφείς διατάξεις, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια δικαίου. Τα έχει τονίσει αυτά και η Εποπτική Επιτροπή. Θεωρούμε ότι χρειάζονται μηχανισμοί που δεν θα επιτρέπουν άσκηση πίεση στον Γενικό Διευθυντή, ούτε και υπέρβαση των ορίων καθηκόντων του. Έχουμε για παράδειγμα και τρέχουσε διαδικασίε κατά επιτρόπων. Θα θέλαμε να μάθουμε τι γίνεται. Ολόκληρε οι Βρυξέλλε μιλούν γι' αυτό και κανεί δεν λέει σε εμά τίποτε. Είναι σημαντικό λοιπόν για το ερώτημα πότε αρχίζει η έρευνα, να υπάρχει υποχρέωση κοινοποίηση και στην Εποπτική Επιτροπή και ιδίω όταν απορρίπτει την έναρξη διοικητικών ερευνών για μια υπόθεση ο Γενικός Διευθυντής. Υπάρχουν 64 υποθέσεις που εκκρεμούν και αναμένουμε τις περαιτέρω πληροφορίες. η συνέχεια που δίνεται στις ε, έρευνες του Όλαφ επίσης είναι ένα θέμα, διότι συχνά οι χώρες μέλη δεν θέλουν ή και δεν μπορούν να δώσουν συνέχεια στις ε, έρευνες, διότι δεν υπάρχει υπαρκής προστασία. Δεν πρέπει ε, να χάσουμε την ευκαιρία εδώ να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό και να ενισχύσουμε και τα διαδικαστικά δικαιώματα Ανησυχώ κύριε Επιτρόπε, διότι τώρα δεν έχουμε δει μελέτη για διοικητικέ έρευνε στι χώρε μέλη. Και τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται να κάνουν οι διοικητικέ αυτέ έρευνε. Εμεί τουλάχιστον δεν τα έχουμε τα στοιχεία αυτά. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο, σα παρακαλώ να μα το διαθέσετε, διότι μπορούμε τότε να διασυνδέσουμε τι δραστηριότητε του Όλαφ καλύτερα με αυτέ των χωρών μελών. Παρακολουθώ τι δράσει του Όλαφ εδώ και 14 χρόνια που είμαι ευρωβουλευτή. Σε ένα πραγματικό δίκιο διαρκούν πάρα πολύ. Υπάρχουν ελλείψεις τις οποίες όμως πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Θέλουμε ο Όλαφ να εκμεταλλευτεί τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελία για να ενισχύσει και τη δική του δραστηριότητα. Βλέπουμε ότι έχουν μειωθεί σημαντικά τα ανακτώμενα ποσά βλέπουμε ότι γίνονται συστάσεις από τον Όλαφ και αυτά τα ποσά αυξάνουν. Αλλά οι πραγματικές ανακτήσεις ποσών μειώνονται. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να σας απασχολήσει και εσάς κύριε Επιτροπέ. Γιατί δεν τα καταφέρνουμε να ανακτήσουμε τα ποσά την οποία συνιστά την ανάκτηση ο Όλαφ. Έχουμε εξετάσει και εμείς την έκθεση και όταν βλέπουμε από την Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης και όχι την πιο πρόσφατη διεύθυνση, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από ορισμένα πράγματα να πάρει ούτε ένα ευρώ από τα διαρθρωτικά ταμεία δηλαδή, να ανακτήσει ούτε ένα ευρώ. Και εν ώψη του πλήθου των υποθέσεων που έχουμε, θεωρώ ότι έχουμε ένα θεμελιώδες πρόβλημα. Το οποίο θεμελιώδες πρόβλημα νομίζω πρέπει κάποτε να μας απασχολήσει. Η πρόσβαση λοιπόν, βεβαίω, τα διαδικαστικά δικαιώματα αποτελούν ένα δύναμο σημείο, και η κριτική που ασκούν πολλοί συνήγοροι περάσπιση ανά την Ευρώπη εστιάζεται εκεί. Δεν είμαι βεβαία ότι μέχρι τη δεύτερη φάση της αναθεώρησης μπορούμε και θα έπρεπε να περιμένουμε. Στο γραφείο μου έρχονται πολλοί και μου μιλούν διότι καταστρέφεται η ύπαρξή τους ως αξιωματούχων και είμαι υποχρεωμένο να του πω αν πρέπει να περιμένετε δύο, τρία, τέσσερα χρόνια. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Και γι' αυτό θα χρειαστεί περαιτέρω επεξεργασία και ελπίζω και το Συμβούλιο να εγκύψει στο θέμα αυτό. Αν και από τι διαβουλεύσει του Συμβούλιο ω τώρα έχω διαπιστώσει ότι δεν ενδιαφέρονται καθόλου οι Υπουργοί. Θέλουμε βεβαίω και η Εποπτική Επιτροπή να έχει διαρκή πρόσβαση στι εκθέσει του Όλαφ τις εκθέσεις δηλαδή που διαβιβάζονται και στις ε, εθνικές αρχές. Γνωρίζουμε τις εξελίξεις των τελευταίων ετών και δεν θέλουμε να τις αποδεχθούμε πλέον. Οι διαδικασίες και σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγγυήσει για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Το έχει πράξει αυτό και η Εποπτική Επιτροπή. Εναλλακτικά θα μπορούσαν να ενισχυθούν οι αρμοδιότητε τη Εποπτική Επιτροπή και να βελτιωθεί η στελέχωσή, τη. Κάποιε προτάσει τη Επιτροπή έχουν αποσυρθεί βέβαια διότι είναι δύσκολο το πρόβλημα. Αν θα μπορέσει να επιληθεί τώρα δεν είμαι βέβαια, αλλά τουλάχιστον θα κάνουμε την προσπάθεια. Χρειάζεται να κοιτάξουμε τις νομικές βάσεις. Υπάρχουν τουλάχιστον τρει νομικές βάσεις, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις χώρε μέλη. Η πρόταση, η νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν αναφέρεται στο θέμα αυτό. Τώρα, προστίθεται μία ακόμη νομική βάση με τον νέο κανονισμό της ε, Ευρωπαϊκής Αγγελίας, άρα το πρόβλημα του κατακαιρματισμού των νομικών βάσεων οξύνεται περισσότερο. Το πρόβλημα αυτό του κατακαιρματισμού πρέπει να λυθεί, τουλάχιστον πρέπει να περιληφθούν οι εσωτερικές διατάξεις, όπως έχει πει η κυρία Γιάλα Σέντερ με τροποποίησεις που έχει καταθέσει πρόσφατα και θεωρούμε ότι τα διαδικαστικά δικαιώματα είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Λυπούμε που μακρηγόρησα κι εγώ και ο Επίτροπο πρέπει να τρέξει τώρα στο Συμβούλιο Υπουργών. Θα ήθελα όμω να δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Κον, που είναι σκιώδη συζητητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσά κύριε Επίτροπε για την παρουσίαση του εγγράφου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι σχετικέ εξηγήσει τις οποίε υποστηρίζω τουλάχιστον σε ένα σημείο, δηλαδή ότι πράγματι θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρξει ένα εύλογο χρονοδιάγραμμα ώστε να διαμορφωθεί σωστά και με νομική ασφάλεια η λειτουργία της ε, Ευρωπαϊκής Εγγελίας που αρχίσει το 2020. Προβλέπονται σημαντικές αλλαγές, τις εξήγησε και η Πρόεδρος και πρέπει να δούμε εάν πράγματι τώρα πρέπει να επιφέρουμε όλες τις αναγκαίες αλλαγές τώρα, σε μία φάση, ή μπορούμε να δεχθούμε την προσέγγιση δύο φάσεων που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνώ επίσης με τα όσα είπατε για τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Ότι χρειάζεται δηλαδή βελτιωμένη ευρωπαϊκή και διακρατική συνεργασία και θα παρακαλέσω τον Επίτροπο να θέσει το θέμα αυτό σήμερα ήδη στο Συμβούλιο Υπουργών, διότι χρειάζεται μεγαλύτερη διαθεσιμότητα και προθυμία από πλευρά χωρών μελών. Δηλαδή, ε, να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που ε, δίνει ο Όλαφ για να διεξάγουν τις σχετικές έρευνες. Και είναι προφανές ότι υπάρχει σημαντικός χώρος βελτιώσεων. Έχω ορισμένε ερωτήσει εν προκειμένου και πρώτα την ερώτηση προ εσά, κυρία Πρόεδρε, πώ βλέπετε το χρονοδιάγραμμα. Αν δηλαδή προβλέψουμε μεγαλύτερη έκταση τροποποίησεων και προ εσά, κύριε Επίτροπε, εάν θέλουμε να ξεκινήσει το 2020 η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τι δραστηριότητε της, πότε θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η κοινοβουλευτική επεξεργασία του κειμένου και πιο συγκεκριμένα ποια θα είναι η συνεργασία Όλαφ και Ευρωπαϊκής Αγγελίας με τις εθνικές αρχές. Διότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν θα έχει εκτελεστικά όργανα. Και επομένως θα πρόκειται για μια διαδικασία όπου θα εμπλέκονται και οι χώρες μέλη και οι χώρες μέλη που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή αγγελία και αυτές που δεν συμμετέχουν. Πώς λοιπόν θα διαμορφωθεί η ασφάλεια δικαίου τώρα για τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Αυτές είναι οι ερωτήσει μου και αναμένω τη συνεργασία μαζί σας. Ο κύριος Κλίντς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η αναθεώρηση του κανονισμού του Όλαφ όντω έχει επίγοντα χαρακτήρα. Προσφέρει και ευκαιρίες αλλά ε, ε, κρύβει και κινδύνους. Κατά τη γνώμη μου ο πολίτης δεν έχει πλήρη κατανόηση για την εργασία, της εργασίας μάλλον του Όλαφ και ούτε γνωρίζει καν ότι ο Όλαφ περιορίζεται στην διαρεύνηση διοικητικών παρατυπιών και για το λόγο αυτό οι πολίτες συχνά είναι απογοητευμένοι. Τώρα με τον παρόντα κανονισμό έχουμε την ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε στους πολίτες ποια είναι η αφετηρία για ποιο λόγο ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τι μπορεί να αναμένει κανεί στο μέλλον από του δύο αυτού φορεί. Γι' αυτό και πρέπει να γίνει η επεξεργασία του κανονισμού, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια ε, στοχευμένη επικοινωνία. Γνωρίζουμε όλοι ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει μεγάλε δυσχέρειε επί του παρόντο και ότι το ευρωπαϊκό εγχείρημα δεν προχωρεί όπω θα θέλαμε. Για να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτε δεν θα ε, απογοητευτούν έτσι περισσότερο, πρέπει να δούμε τι ακριβώς μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που οι πολίτες θεωρούν ότι λείπει είναι ότι δεν μπορούν, μπορούν να αντιληφθούν ότι όλα δεν είναι εισαγγελική αρχή. Και γι' αυτό οι πολίτες όταν μαθαίνουν για παρατυπίες ή και για εγκληματικές υποθέσεις δεν κατανοούν γιατί γίνεται απολύτως τίποτε συγκεκριμένο. Και γι' αυτό λοιπόν είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει, να υπάρξει επικοινωνία και διευκρίνηση. Η στόχη τώρα της ε, ε, αναθεώρησης του κειμένου είναι ξεκάθαρη. Ότι θα πρέπει να είναι μια διαδικασία σε δύο φάσεις, μου φαίνεται εν ώψη του γεγονότος ότι η κοινοβουλευτική θητεία λύγει σε λιγότερο από ένα χρόνο, μου φαίνεται λογικό. Όμως είναι κρίσιμο ήδη τώρα να είναι σαφές Προ τα που κατευθυνόμαστε. Και εδώ προκύπτει για μένα μια ερώτηση, διότι για την ώρα φαίνεται σαν να είναι όλα ξεκάθαρα. Διατηρούμε τον Όλαφ ως ισότιμο εταίρο, όπως είπε και ο επίτροπο, ισότιμο εταίρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελία και ιδρύουμε εξ αρχή την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αν όμω, δεν πούμε ξεκάθαρα στου πολίτε ποια είναι η αφετηρία, δεν θα είναι για τους πολίτες τίποτε άλλο παρά η δημιουργία ενός ακόμη οργανισμού. Δηλαδή θα πούν οι άνθρωποι δεν τους φτάνει πια ό,τι έχουν στις Βρυξέλλες, όλα αυτά που έχουν φτιάχνουν άλλον οργανισμό. Γι' αυτό και είναι απαραίτητο να καταστεί σαφές ότι δεν πρόκειται μόνο για νέα αρχή η οποία θα έχει νέα καθήκοντα, αλλά ότι είναι και μια αρχή την οποία χρειαζόμαστε απαραίτητα. Και εκεί θα πρέπει να παίξουν τον ρόλο τους και οι χώρες μέλη. Γι' αυτό για μένα τίθεται το ερώτημα εάν μακροπρόθεσμα όταν θα μπούμε στη δεύτερη φάση δηλαδή, αν χρειαζόμαστε όντως δύο φορείς, Όλαφ και η ή αν θα πρέπει από τώρα να εργαστούμε πάνω σε μια συγχώνευση των δύο φορέων, διότι σε πολλές χώρες μέλη υπάρχουν ε, αρχές οι οποίες κάνουν και τα δύο, δηλαδή και τις διοικητικές έρευνες και την ποινική δίωξη υπό μία στέγη για τον πολίτη δεν είναι κατανοητό ότι ο Όλαφ ξεκινά και διεξάγει έναν αριθμό ερευνών, στο τέλος όμως δεν καταλήγει πουθενά. Δεν καταλαβαίνει ο πολίτης ότι ζητούνται ανακτήσεις, αλλά ποτέ στην πραγματικότητα δεν ανακτάται ούτε ένα λεπτό του ευρώ. Αν τα πράγματα αυτά δεν αλλάξουν, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την απογοήτευση πολλών Ευρωπαίων πολιτών Αντίθετα, ρίχνουμε νερό στον μήλο των λαϊκιστών, οι οποίοι ευχαρίστως χρησιμοποιούν τέτοια επιχειρήματα για να γκρεμίσουν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Ξαναλέω λοιπόν, οι προσδοκίε των πολιτών μπορούν να επηρεαστούν θετικά με την παρούσα τροποποίηση του κανονισμού, αλλά πρέπει να την ξεκινήσουμε σωστά. Πρώτα-πρώτα πρέπει να φροντίσουμε τα δικαιώματα του ατόμου να είναι προστατευμένα στις διαδικασίες αυτές. Να μην κατηγορήσουν ότι με καλές μεν προθέσεις προχωρούμε σε τροποποίησεις, αλλά ξεχνούμε τα δικαιώματα, τα διαδικαστικά δικαιώματα των ε, ε, ατόμων. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα τα είπατε εσείς όλα. Όταν ακούω τα όσα λέει εδώ η πρόεδρός μας για το χρονοδιάγραμμα, μας μίλησε προηγουμένως για 14 χρόνια που παρακολουθεί το, τις του Όλαφ. Εγώ είμαι μία μόνο ένα χρόνο εδώ μέλος και ήδη έχω να σπίσει τα μαλλιά μου από αυτά που βλέπω εδώ, αλλά θεωρώ πάντως ότι όλα αυτά που μου προτείνετε είναι σκόπιμα και θετικά, υπάρχουν όμως όπως εξήγησα και ευκαιρίες και κίνδυνοι και αν δεν τα καταφέρουμε καλά θα προσθέσουμε και άλλη απογοήτευση σε αυτήν που αισθάνονται οι πολίτες. Πρόεδρος, έχω άλλους δύο συναδέλφους. Σας παρακαλώ όμως περιοριστείτε σε δύο λεπτά ο καθένας. Η κυρία Γιάλα πρώτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας και για το έγγραφο εργασίας. Μας παρουσιάζετε εδώ κάποια θέματα και φυσικά ε, συμφωνούμε με τις ανησυχίες αυτής της Επιτροπής Επίσης, ε, συμφωνώ με την ανησυχία ότι δεν ε, εκμεταλλευόμαστε επαρκώς την ευκαιρία αναθεώρησης του κανονισμού της όλα αυτή τη στιγμή που πρέπει να ενισχύσουμε την ε, πολύπλοκη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, χωρίς να δημιουργήσουμε περαιτέρω εμπόδια. Θα ήθελα λοιπόν ο κύριος Έιτινγκερ, καθώς τον άκουσα να μιλά για έναν εταίρο με πλήρη δικαιώματα. Θα ήθελα να μου πει αν η Κομισιόν θα μας ε, πει ξεκάθαρα ποια θα είναι η απαραίτητη ιεράρχηση μεταξύ των δύο υπηρεσιών. Γιατί διαφορετικά αρχίζουμε από την αρχή να δημιουργούμε γκρίζε ζώνε και αν κανείς δεν ξέρει ποιος θα κάνει τι, είναι σίγουρο ότι θα ξεκινήσουν διάφοροι διαξυφισμοί για το ποιος θα αναλάβει τι. Και μπορεί να γίνει πολύ πολύπλοκη κατάσταση. Εγώ θα προτιμούσα να ενισχύσουμε και να βελτιώσουμε τα διοικητικά καθήκοντα όπου πρέπει να επικεντρωθεί η Όλαφ και αυτό πρέπει να γίνει με τη μεγαλύτερη δυνατή λεπτομέρεια και να παραμείνει πολύ ξεκάθαρο η αυτή η ιεράρχηση. Διαφορετικά θα έχουμε αυτές τις γκρίνες ζώνες. Και όπως ε, είπε και η συγχύτρια, υπάρχει και το πρόβλημα των δικονομικών εγγυήσεων ε, και υπάρχει και το περίφημο εγχειστήριο. Οπότε δεν μπορέσαμε να βρούμε την κατάλληλη βάση και να το εντάξουμε με έναν κατάλληλο τρόπο. Έτσι λοιπόν ε, τελικά παράγονται καταστάσεις όπου είδαμε και στο παρελθόν όπου η ανεξαρτησία της Όλαφ είχε τεθεί υπομφισβήτηση. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν για το θέμα των εγγυήσεων. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα γίνει. Εγώ θα προτιμούσα να βελτιώσουμε τις δράσεις της Εποπτικής Επιτροπής. Θα το δούμε και όταν ο κύριο Μούλτερ μας παρουσιάσει την έκθεσή του. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πράξουμε έτσι ώστε και η Εποπτική Επιτροπή να ενισχυθεί για να μπορεί να διαφυλάσει τις δικονομικές εγγυήσεις και την ανεξαρτησία της όλων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αλαφράγκα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Να πω ότι και εμείς ε, θεωρούμε ότι είναι πολύ πλοκό το θέμα. Η θέση σε σχέση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ε, μας δίνει την ευκαιρία να λύσουμε το ε, νομικό πλαίσιο που δεν είναι ξεκάθαρο ως προς τη λειτουργία της Όλαφ και έχουμε λοιπόν μια ιδιαίτερα κατάλληλη ευκαιρία για να προσπαθήσουμε να λύσουμε τα προβλήματα που έχουμε επιτάπητος στο πλαίσιο αυτό, Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει κάτι θεμελιώδες και συνίσταται στο να δούμε, να ξέρουμε ποια είναι η φύση που θέλουμε να έχει όλα. Εγώ νομίζω ότι αυτό το εξηγείται πολύ καλά στο έγγραφο εργασία. Αν θέλουμε μια αυτόνομη υπηρεσία που θα είναι αρμόδια για τι διοικητικέ έρευνε, για όλα τα ζητήματα που μπορούν να βλάψουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης ή αν θέλουμε να λειτουργεί ως προσάρτημα η Όλαφ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Υπό την έννοια αυτή, τα εκκρεμή ζητήματα για τις εσωτερικές έρευνες, για τις εξωτερικές έρευνες, για τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη, για τα θέματα των εγγυήσεων ε, των ε, υποκειμένων των ερευνών, θα πρέπει να βρίσκονται στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας. Νομίζω ότι είναι εξαιρετική ευκαιρία. Το έγγραφο εργασία καλύπτει όλα τα στοιχεία επί των οποίων εμείς θα πρέπει να τοποθετηθούμε και με άλλους νομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι είναι εξαιρετική ευκαιρία για να προσπαθήσουμε να βάλουμε τάξη και να καταρτήσουμε με ε, σαφήνεια Ποιε είναι οι αρμοδιότητε των δύο οργανισμών. Θα πρέπει να αποφύγουμε τι επικαλύψει. Δεν μπορούμε ε, να μπούμε εδώ σε ε, μία διένεξη για τι αρμοδιότητε. Έτσι λοιπόν έχουμε τώρα την ευκαιρία να αποσαφηνίσουμε πώς οι οργανισμοί αυτοί θα υπηρετούν τις έρευνες στον ποινικό και στο διοικητικό τομέα για να υποστηρίξουν και να περασπίσουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ενδιαφέρει βέβαια και το θέμα του χρόνου Κάποια στιγμή θα πρέπει να τοποθετηθούμε για τις προτάσεις της Κομισιόν και νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τη συζήτησή της για τη φύση των οργάνων που είναι συζήτηση αυτή τη στιγμή και επί των νομοθετικών προτάσεων που μας παρουσιάζει η Κομισιόν. Ευχαριστώ. Εσείς κύριε Επιτροπή, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις σας, τις οποίες βρίσκω απολύτως ε, λογικές και αντικειμενικές και τις προτάσεις και τις προσδοκίες σας. Σε ό,τι αφορά την οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων, πρέπει να εξετάσει κανείς πώς θα αποφύγει την διαφωνία ή, εν πάση περιπτώσει, τις ασάφειες και την σύγκρουση αρμοδιοτήτων στο μέλλον. Για μένα είναι ξεκάθαρο ότι με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχωρούμε σε ένα τομέα, τον εθνικό, περιφερειακό, τοπικό, που δεν υπάρχει από την αρχή της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία ιδρύθηκε με πρώτα μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βεβαίως το Συμβούλιο και αργότερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά η εκτέλεση ποτέ δεν έγινε μέσω Ευρωπαίων αξιωματούχων. Είχαμε λοιπόν αφενό προπολογισμό από εκεί τι πληρωμέ, κάτι έπαιρνε ο Γιώργος. εν τέλει, από την άλλη μεριά η πολιτική τη συνοχή με επιμερισμένη διαχείριση, κοινή διαχείριση. Έχουμε μια συνθήκη, είναι σαφή η ρόλη εκεί των κυβερνήσεων, υπουργείων, περιφερειών κλπ. Και κατά βάση αυτό που ήμασταν εμείς ήμασταν ένα είδος γραμματείας, ένα είδος ε, ταμείου πληρωμών. Και γι' αυτό οι χώρες μέλη προτιμούν οδηγίες και όχι κανονισμούς για να μπορούν να αποφασίζουν οι ίδιες πώς και τι και πότε το κάνουν. Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν περισσότεροι κανονισμοί, δηλαδή άμεσα εφαρμοστέο ευρωπαϊκό δίκαιο και η τάση είναι τώρα να είναι και η εκτέλεση στα χέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους σύγχρονους ευρωπαϊκούς προπολογισμού υπάρχουν και προγράμματα Όπω ε, η διευκόλυνση συνδέοντα την Ευρώπη, όπου εμεί αποφασίζουμε το ευρωπαϊκό επίπεδο δηλαδή ποιε είναι οι προτεραιότητε. Βλέπετε την διόρυγα του Μπρένερο και αλλού. Εμείς, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τα τελευταία χρόνια δηλαδή έχουμε επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πλησιάσει περισσότερο τα έργα, περισσότερο να φτάσει κοντύτερα στον δικαιούχο δηλαδή των πληρωμών. Μέχρι τώρα για την καταπολέμηση των παρατυπιών και των απατών όταν πρόκειται για έργα εκτός Βρυξελών επαφιέμεθα στην συνεργασία των εθνικών, περιφερειακών, τοπικών επιπέδων σε ό,τι αφορά παρατυπίες για, τους, ε, για τον εσωτερικό μας οργανισμό, για τους δικούς μας αξιωματούχους δηλαδή, είμαστε εμείς άμεσα αρμόδιοι. Όμως για παρατυπίες σε έργα συνοχής, σε έργα διαρθρωτικά, στο, σε μέγιστο βαθμό εξαρτώμεθα τότε από τις εθνικές και περιφερειακές αρχές, και τις εθνικές εισαγγελίες. 28 χώρες μέλη και 280 ξεχωριστές περιφέρειες δεν δρούν βεβαίως και δεν μπορεί κανείς να το παραγνωρίσει αυτό με τον ίδιο τρόπο. 28 που είναι όλοι ίσοι αλλά όχι όλοι ίδιοι. Κάποιοι είναι καλύτεροι σε ένα τομέα, άλλοι σε έναν άλλο. Ποτέ όμως δεν είναι οι ίδιοι πάντοτε παντού καλύτεροι. Εκτός από τους δύο Ισπανούς ευρωβουλευτές, άκουσα μόνο γερμανικά μέχρι τώρα προσοχή ε, κρότο κόδωνα του κινδύνου να μην υπάρξει ένα είδος γερμανικής αλαζονίας, το οποίο δεν θα εξυπηρετήσει κανένα. Δηλαδή, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι πρώτον υπάρχουν νέε χώρε μέλη, οι οποίες χρειάζονται κάποια χρόνια ακόμη εξέλιξη και ανάπτυξης μιας νοοτροπίας που να ανταποκρίνεται στου δημοκρατικού κανόνε διαφάνεια. Αυτό αφορά βεβαίω όχι μόνο νέε χώρε, αλλά και παλέ χώρε μέλη. Που καμιά φορά υπάρχουν και πόνοι συγκάλυψη και όχι ε, απόλυτη διαφάνεια. Εμεί, σε ό,τι αφορά την φιλοσοφία και την προσέγγιση μα, βασιζόμαστε στη συνεργασία των δύο φορέων, η Ευρωπαϊκή Αγγελία και όλα και όχι άκαμπτη διάκριση των αρμοδιοτήτων των μεν και των δε. Βέβαια, η πράξη θα τα δείξει αυτά. Ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Αγγελίας σε συνεργασία με τον διευθυντή του Όλαφ και βεβαίως και, η επιχειρησιακή, και το επιχειρησιακό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε μετά από δύο ή τρία χρόνια της δραστηριότητας μετά από 2-3 χρόνια να δούμε αν χρειάζεται πράγματι περισσότερη διάκριση ακόμη ή εάν μπορεί να ε, καταδείξει την αξία της μια συνεργασία. Βεβαίω φαιές ζώνες θα υπάρχουν παντού. Γνωρίζω ήδη πολλές φαιές ζώνες και μεταξύ γενικών διευθυντών, γενικών διευθύνσεων. Ακόμα και μεταξύ επιτρόπων. Εάν προλάβει ο Α επίτροπος πιο γρήγορα από κάποιον άλλον μπορεί να πάρει αυτό σε ένα θέμα. Τα ίδια ακούω ότι υπάρχουν και στο Κοινοβούλιο, συγκρούσει αρμοδιοτήτων δηλαδή μεταξύ κοινοβουλευτικών επιτροπών. Έχω καταστεί μάρτη και συζητήσεων σχετικά με το ποια είναι η αρμόδια επί τη ουσία κοινοβουλευτική επιτροπή όταν έχετε μια πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα αναλάβει η Επιτροπή ε, ε, Δικαιοσύνη ή άλλη επιτροπή, η Επιτροπή Βιομηχανία ή η Επιτροπή Περιβάλλοντο. Και αυτό καμιά φορά είναι ανοιχτό ως θέμα. Όλοι έχουμε μια εμπειρία στον κόσμο αυτό. Εάν δηλαδή προσπαθήσουμε να βάλουμε ήδη από τώρα στο νόμο ζητήματα σύγκρουση αρμοδιότητας που μπορεί να προκύψουν σε πέντε χρόνια, αυτό δεν μπορεί να γίνει από τώρα. Θα πρέπει να αναμένουμε συνεργασία των δύο αυτών υπηρεσιών. Να προβλέψουμε τη συνεργασία, παρόλα αυτά να επιτρέψουμε ταυτόχρονα και την διάκριση των αρμοδιοτήτων. Εμένα, στο χαρτοφυλάκιο, με ενδιαφέρει η σταθεροποίηση του Όλαφ. Δηλαδή, η ίδρυση τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην αποβεί ει βάρο του Όλαφ, ούτε σε ό,τι αφορά τη στελέχωση, δηλαδή με αφαίρεση θέσεων οργανογράμματο, αυτό νομίζω ότι έχει επιληθεί δικαίω, ούτε ε, στην χρηματοδότησή του, ούτε στην νομική του βάση. Και επομένω στην βάση που θα επιτρέπει την λειτουργία του. Δεν θα τροποποιήσουμε πλέον εμείς τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Δεν επηρεάζουμε δηλαδή τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Αγγελίας με τα προβλεπόμενα στην αναθεώρηση του κανονισμού του Όλαφ. Ο νέος κανονισμός, ΕΠΟ δηλαδή, θα παραμείνει ως έχει, με, όλες, με όλα τα ισχυρά σημεία που έχει και ίσως και με κάποιες αδυναμίες. Θα σας παρακαλέσω τώρα που θα έρθει νέος Γενικός Διευθυντής και είδαμε και ο εκτελών καθήκοντα Γενικού Διευθυντού θεωρώ ότι έκανε πάρα πολύ καλά τα καθήκοντά του, δώστε στον Γενικό Διευθυντή του Όλαφ επαρκή περιθώρια διαχείριση των υποθέσεων. Ποια υπόθεση θα, ε, υπόθεση θα επιληφθεί, ποια θα αποφασίσει να μην επιληφθεί. Ο έλεγχος του Γενικού Διευθυντού του Όλαφ είναι σωστός, αλλά θα πρέπει να είναι γενικός διευθυντή και όχι ένα είδος γενικού γραμματέα που ελέγχεται δηλαδή διαρκώ. Κατά βάση μεταξύ εισαγγελία και Όλαφ, από τη μια μεριά ποινική δίωξη, από την άλλη μεριά προστασία των οικονομικών συμφερόντων. Αυτοί είναι οι δύο μεγάλοι στόχοι. Ποινική δίωξη σημαίνει εισαγγελία, προστασία των ε, οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κυρίως Όλαφ. Ασκείται κριτική σχετικά ότι δεν γνωρίζετε, σχετικά με το ότι δεν γνωρίζετε αρκετά σχετικά με τα ανακτώμενα ποσά. Ο Όλαφ κάνει την προεργασία και καταλήγει σε συστάσεις. Η ανάκτηση επιτόπου δεν είναι υπόθεση του Όλαφ. Ο Όλαφ δεν είναι δικαστικός επιμελητής. Αυτά οφείλουν να τα κάνουν οι γενικέ διευθύνσει. Μπορεί να ελέγξει κανεί αν μια γενική διεύθυνση τα καταφέρνει καλύτερα από μια άλλη. Αλλά η Γενική Διεύθυνση Έρευνα και Ανάπτυξη, για παράδειγμα, ε, η ψηφιακή ή των προπολογισμών, κινητοποιούνται στην βάση των συστάσεων του Όλαφ και αυτές είναι οι υπεύθυνε για την επίτευξη της ανάκτησης των καταβληθέτε των ποσών. Μιλήσατε και για την προθεσμία των 30 ημερών. Δεν είναι όμως αποκλειστική η προθεσμία αυτή. Η ΕΠΟ θα πρέπει να πει μετά από 30 ημέρες, ναι, επιλαμβανόμαστε τις υπόθεσεις. Μπορεί όμως και μετά από τις 30 ημέρες να το δηλώσει αυτό. Δηλαδή, πρόκειται για μια προθεσμία, για μια πρώτη τοποθέτηση. Δεν είναι όμως αποκλειστική η προθεσμία αυτή διότι προβλέπεται και μετά άλλη τριακονθήμερη προθεσμία για δραστηριοποίηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τελειώνοντας, δύο σχόλια. Πριν από το τέλος της κοινοβουλευτικής αστήτειας, θα ήθελα να μου δώσετε μία λίστα, ένα κατάλογο ελήψεων, ένα κατάλογο ε, πραγμάτων που θέλετε να αναθεωρηθούν και να μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει την υποχρέωση σε ένα χρόνο, στη δεύτερη φάση δηλαδή, να υποβάλει τη νέα, το νέο σχέδιο τροποποίησης και εκεί να μπορείτε να πείτε εσείς ναι, όχι, να υποβάλλετε δηλαδή τον κατάλογο των πραγμάτων που αναμένετε να κάνουμε, τις προσδοκίες σας. Δεύτερο, για το θέμα της ενίας νομικής βάσης δεν θα προλάβουμε τώρα, θα μπορούμε όμω να προσφέρουμε και ψηφιακά και επί χάρτου να σας υποβάλουμε ένα κομπέντιουμ όπου θα περιλαμβάνονται όλες οι νομικές βάσεις, όλα τα νομοθετήματα, όλες οι παράγραφοι σε έτερα νομοθετήματα τα οποία αφορούν την δράση του Όλαφ. Αυτά μπορούμε να τα έχουμε στη διάθεσή σας μέχρι την άνοιξη του επόμενου έτους. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, αντιλαμβάνομαι ότι, ότι ε, πρέπει να φύγετε, αλλά έχω την ερώτηση του κυρίου Κον, το χρονοδιάγραμμα. Το χρονοδιάγραμμα δεν μπορεί να αλλάξει. Υπάρχει πίεση χρόνου λόγω της ίδρυσης της ε, Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Αποτελεί πίεση διότι το Συμβούλιο είναι εκείνο το οποίο δεν θα επιτρέψει να προχωρήσει. Θα μας υποσχεθεί τα πάντα αλλά σας ξαναθυμίζω, η προηγούμενη τροποποίηση του κανονισμού όλα χρειάστηκε πέντε χρόνια και δεν ήταν δική μα η καθυστέρηση. Υπάρχει λοιπόν πίεση χρόνου, όντω, ε, υπάρχει κίνηση και αυτό θα μας επιτρέψει να εξαλείψουμε κάποιες βασικές ελλείψεις τις οποίες ε, δεν διορθώνει δυστυχώς η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι και ζητήματα, ε, ευαίσθητα νομικά ζητήματα, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να μπορέσουμε να επιλύσουμε. Λυπούμε πολύ που ε, μιλούν μόνο Γερμανοί ευρωβουλευτέ πράγματι εδώ. Είμαι ευγνώμων στου δύο Ισπανού ευρωβουλευτέ, αλλά εν πάση περιπτώσει μου φαίνεται ότι πάντα οι ίδιοι είναι παρόντε και παρούσε εδώ. Δεν έχει σχέση με αλαζονία, ούτε δεν ξέρω αν έχει σχέση με αλαζονία ή με Κουταμάρα. Εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι η απάλληψη επικαλύψεων αρμοδιοτήτων είναι κάτι που αξίζει τον κόπο. Πόσο χρόνο περνάτε για να αντιμετωπίσετε επικαλύψεις αρμοδιοτήτων. Το ίδιο και εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά πρέπει να φροντίσουμε να αρθούν εκ των προτέρων μέσα από τα ίδια τα νομοθετήματα. Να είναι σαφές ότι ο Α κάνει Αυτά τα πράγματα ο Β' κάνει τα άλλα πράγματα. Μπορεί να είναι διασκεδαστική καμιά φορά η σύγκρουση αρμοδιοτήτων, αλλά δεν θέλουμε να υπάρχει. Θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μπορέσει να λειτουργήσει. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά σα, τα καθήκοντά τη. Διότι αλλιώ προκαλούμε αυτό που λέει ο κ. Κρίν. Δηλαδή απογοήτευση, διότι θα φτιάξουμε άλλη μια αρχή η οποία πάλι δεν θα μπορεί να εκτελήσει τα καθήκοντά τη. Κύριε Επίτροπε, αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να φύγετε, αλλά αν δει κανεί τον Όλαφ, ναι, μεν έχουν γίνει πολλά πράγματα, αλλά 20 χρόνια υπάρχει ε, Όλαφ και εξακολουθεί να έχει ανάγκη μεγάλων βελτιώσεων. Μια ερώτηση που νομίζω πρέπει να την θέσει η σε αυτήν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμεί είμαστε το επικοδομητικό τμήμα της σύνομοθετική διαδικασίας αμέσως μετά τις ελληνές διακοπές, εγώ θα ρίξω όλο μου το βάρος στη διαδικασία αυτή, διότι εμείς θέλω να αποδείξουμε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλαδή, είμαστε μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλές διακοπές κύριε Επίτροπε. Προχωρούμε αμέσω στο επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως που είναι το υπαριθμό 13 παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης της Όλαφ, του Όλαφ για το 2017. Κύριε Άιλετ, δεν μπορέσαμε να έρθουμε ή δεν θα μπορέσουμε να έρθουμε στο πάρτι που θα οργανώσετε. Βλέπετε όμω είναι και δύσκολο να ε, επιτύχω να προσέλθουν οι ευρωβουλευτέ καν εδώ στην ε, συνεδρίαση. Να σα δώσω πολύ ευχαρίστω τον λόγο για την παρουσίαση τη ετήσια έκθεση ε, του Όλαφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και συγχωρήστε με. Δεν είναι απόλυψη σεβασμού που το άργησα, αλλά επειδή επιφυλάχθηκα όσον αφορά την κυκλοφορία του Προέδρου Τραμπ, πήρα το μετρό, τέλο πάντων, ε, για να μην μπλοκαριστώ, τελείως άργησα. Για να δούμε τώρα την ετήσια έκθεση ε, για την Όλαφ. Ευθύς να σας πω ότι επί 10 μήνες είχαμε τον Τζοβάνι Κέσλερ στο τιμόνι και εκείνος θα πρέπει να πιστωθεί και όχι εγώ τα εκεί επιτέμματα. Α, βεβαίως θα πρέπει να πούμε μπράβο και στο προσωπικό της υπηρεσίας χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν να έχουμε τόσες επιτυχίες ε, και βεβαίως επισημαίνουμε και πάλι όλες αυτές τις δυσκολίες που συναντήσαμε για να δούμε τώρα τα της έκθεσης. Να δούμε. Ε, δεν μπορώ να σας ε, πω ε, ε κάποιο γενική εποπτεία όλων των, των α, δραστηριοτήτων γιατί έχουμε εδώ στατιστικά, έχουμε πάρα πολλά αλλά τα τελευταία χρόνια έχουμε επικεντρώσει την προσοχή μας σε κάποια πιο σημαντικά για να βελτιωθεί η στρατηγική της επικοινωνίας και για να μπορέσουμε τα σημαντικά να τα καταστήσουμε κατανοητά. Οπότε, για να δούμε τώρα τα θέματα του εισοδήματο περισσότερα από τα της δαπάνησαν και το αντίστροφο <laughs> είναι η αλογία στην δουλειά μας. Πάντως, ό,τι θέλετε να σας εξηγήσω για τη δουλειά μας, ευχαρίστως είτε έχετε κάτι να ρωτήσετε από την παρουσίαση, είτε εκτός αυτής. Εδώ εστιαζόμαστε σε μεγάλες διεθνείς υποθέσεις και ελπίζουμε ότι η πυρογνωμοσύνη μας μπορεί να κάνει τη διαφορά υπέρ των φορολογουμένων και έχουμε συστάσεις διατυπώσει που είναι πάνω από 300 συνολικά και έχουμε συστήσει την ανάκτηση τριών δις ευρώ και παραπάνω. Αυτό είναι το ποσό. Αυτό δεν γίνεται συχνά και δεν ξέρω και αν θα ξαναγίνει γιατί ε, απορρέει από κάποιες περιπτώσεις απάντες που συνέτρεξαν και όπως ξέρετε είχαμε και πηγή του Ηνωμένου Βασίλειου και άλλες χώρες και έτσι καταλήξαμε σε αυτή την ανάκτηση. Είχαμε 1.100 επιλογές και 215 έρευνες, 197 έρευνες ολοκληρώθηκαν και άνοιξαν, 215 ξεκίνησαν. Όλα αυτά όσον αφορά την προστασία του προϋπολογισμού από την απάτη. Θεωρήσαμε ότι αυτό είναι η καταξοχή που προσφέρουμε στον Ευρωπαίο συμπολίτη. Για να δούμε τώρα να καταλάβετε καλύτερα την ουσία του έργου μας. Ε, ό,τι, ό,τι ελέγχθη σήμερα το αστεριζόμαστε όλα αυτά γιατί πάντοτε εμείς προσπαθούμε να βελτιωθούμε και δεν είναι πάντοτε εύκολο λόγω των νομικών συνέπειων. Ιδίω όσον αφορά τι έρευνε για τις δαπάνες. Πάντως κάνουμε ό,τι μπορούμε στα πλαίσια των δυνατοτήτων επικοινωνία. Και με αυτή την έκθεση θέλουμε να σας δείξουμε τι ερευνητική δουλειά κάνουμε για να δείτε ποιες είναι οι κυριαρχές τάσεις για τις έρευνες σε σχέση με τα ε, στοιχεία, ενδείξεις, αποδείξεις που έχουμε από τις ε, ολοκληρωθήσεις έρευνες του 17. Άρα, συνεχίζουμε και έχουμε σαν βασικές τάσεις φαινόμενα τη σύγκρουση συμφερόντων, την διαφθορά. Α, ε, βέβαια, το, η σύγκρουση των συμφερόντων είναι μια ενία που θα πρέπει να γίνει περισσότερο κατανοητή. Επίσης, την χειραγώγηση και ατασταλίες σε σχέση με ε, δημόσιους διαγωνισμού, γιατί έχουμε περιπτώσεις όπου το οργανωμένο έγκλημα ε, εκεί στοχεύει για να κερδίσει. Και ε, περισσότερα χρήματα τώρα δαπανώνται για τους πρόσφυγες. Οπότε και οι απαταιώνες ελκύονται από όλα αυτά, οπότε και εμείς αφιερώσαμε χρόνο πολύ για να το αντιμετωπίσουμε. και από πλευράς του μετόπου των τελωνιακών θεμάτων και εκεί έχουμε το διεθνές έγκλημα ε, προς αποφυγή των ε, δασμών και θα επανέλθω σε αυτό το θέμα σε λίγο. Τώρα, για να δούμε κάτι πιο ελαφρύ. Έχουμε εδώ μια υπόθεση που αφορά μικρότερα ποσά, 1,4 εκατομμύρια, όσον αφορά αυτή την έρευνα που είναι σε διάφορα κράτη-μέλη. Ονομάζεται επιχείρηση Χάρτινο Πύργο, Χάρτινο Κάστρο. Συνεργαστήκαμε με τους συναδέλφους στην Ιταλική Οικονομική Αστυνομία, την Guardia di Finanza. προσώπου των οποίων έχουμε σήμερα εδώ κοντά μας και υπήρχε ένας υπερχηματικός όμιλος, ένα κονσότσιουμ το οποίο είχε έδρα την Ιταλία αλλά είναι δραστηριότητες και στη Γαλλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο ούτως ώστε να ελκύουν πόρους για να φτιάξουν ένα νέο τύπου hovercraft το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση θεομηνιών αλλά τελικά αυτό το Hovercraft ποτέ δεν υπήρξε. Και θυμάμαι πριν 50 χρόνια που ήμουν στο σχολείο, είχαμε ναυπηγήσει ένα Hovercraft το οποίο δούλευε. Καλά πήγαινε προς τα πίσω, αλλά τελικά το συγκεκριμένο δεν πήγαινε ούτε μπρο ούτε πίσω. Οπότε έπρεπε τώρα να καθαρίσουμε 12.000 συναλλαγές, να κάνουμε Ελέγχου η Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, σε συνεργασία με τις τοπικέ διοικητικές αρχές τις δύο χώρες και τελικά αυτό που έγινε προσπαθούσαν με πλασταδημολόγια, πλασ... ψεύτικες δαπάνες, με συνεργάτες που ήταν ανύπαρκτοι να πάρουν και άλλα χρήματα. προσπαθούσαν τέλο πάντων να επεξερέσουν τα σχετικά χρήματα με αυτή την απάτη και έτσι να ξεπληρώσουν την υποθήκη για ένα πολυτελές εξοχικό στην Ιταλία. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε εκεί για να ανακτηθούν τα σχετικά χρήματα. Τώρα αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον δεν είναι το ποσό αυτό που όπως είπαμε ε, την κλίμακα των διευθυντικών ταμείων είναι μάλλον μικρό. Απλώ σα τα λέω αυτά για να δείτε ότι θα πρέπει κανεί να μετέρχεται ό,τι μέσο έχει. Ούτω ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει το διασυνοριακό έγκλημα, διασυνοριακή απάτη ε, κατά των κοινοτικών χρημάτων. Αυτά ήταν κάτι σαν για να ξαναγυρίσουμε τώρα στα θέματα των ε, ε, εσόδων. Εδώ βλέπετε τι έγινε αυτές τις περιπτώσεις της απάντησης υποτίμησης ε, εδώ αφορούσε αυτό κάποιες εισαγωγές στο Αμβούργο ε, και η απάτη αφορούσε την εκτελώνηση αυτών των ε, υποδημάτων και κλωστεφαντουργικών και αφορούσε επίσης και η Ηνωμένο Βασίλειο, Σλοβακία, Τσεχία, Γαλλία και Μάλτα. Άλλαξαν αυτοί το σχέδιό τους, οι απαταιώνε γιατί ήταν καλά ενημερωμένοι και ξέρανε πώς να κινηθούν με τα εμπορεύματά τους, όποτε υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Συνεχίζεται το πρόβλημα και τώρα αυτοί οι απαταιώνε ψάχνουν νέα κόλπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι καινούργια κόλπα πάντως και ε, θα έπρεπε να μας έχουν απασχολήσει περισσότερο. Πάντως ε, ήταν αυτά τα εμπορεύματα χαμηλής αξίας, αλλά οι ποσότητες πάρα πολύ μεγάλες. Ο ε, κλασική να είναι τα τσιγάρα, τα οποία δεν πιάνουν πολύ χώρο. Οπότε και εμείς το έχουμε επισημάνει σε όλους τους εμπλεκομένους ότι πρέπει να προσέξουμε αυτά τα φτηνά εμπορεύματα. Μέσω του Αμβουργού λοιπόν νομίζανε οι πατιώνες ότι μπορούν να τη γλιτώσουν και τα κράτη-μέλη προσπάθησαν να επιληφθούν γρήγορα, Μάλτα, Γαλλία και Τσεχία. Οπότε φέτος από ό,τι ξέρουμε, οι επαντιώνες έχουν σταματήσει τα ιστοριότητά τους, τέλο πάντων την έχουν μειώσει και ψάχνουν να δουν από πού αλλού μπορούν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να δούμε τώρα ένα άλλο προϊόν, ένα άλλο εμπόρευμα, μια άλλη πιο μεγάλη απειλή που είναι η δασμία την dumping. Έχουμε θέματα υψηλή τεχνολογία και έχουμε του σχετικού δασμού που επιβάλλονται στου Κινέζου παραγωγού. Εδώ δεν έχουμε εισόδημα το οποίο προκύπτει. αλλά το θέμα είναι η προστασία κατά του αθεμήτου ανταγωνισμού. Και μόλις τις πιστούν οι σχετικοί κανόνες είναι καθήκον μας να τους εφαρμόσουμε. Πολλές φορές ε, τα κυκλώματα του νομίμου εμπορίου μας ενημερώνουν. Πολλές φορές οι Κινέζοι ε, δηλώνουν ότι είναι από την Ταϊβάν ή από την Ιαπωνία. Αυτά τα πάνελ, τα ηλιακά πάνελ, δηλώνεται ότι είναι από αυτές τις χώρες ψευδός και έχουμε ε, συνεργαστεί με στουρανικές αρχές από Βέλγιο, κάτω χώρες και Γαλλία αλλά και Ταϊβάν. Οπότε βλέπετε πόσο είναι απαραίτητο να συνεργαστούμε με τις τελωνικές αρχές και στην Αποανατολή. Πολύ βοήθησε και η συνεργασία με το Βέλγιο, εκτός από την Ταϊβάν. Εννέα είναι οι έρευνε που έχουν ολοκληρωθεί και διατυπώθηκαν για 200 εκατομμύρια ευρώ κάποιες συστάσει. Να, γι' αυτό σας είπα ότι αυτά δύο δίστα, τα οποία εξοικονομήθηκαν από την υπόθεση που αφορούσε το Βασίλειο ήταν κάτι το εξαιρετικό αυτά. Ήδη συζητήσαμε σήμερα τα των ε, συστάσεων και ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι το ζήτημα. Μια που ε, ευθύς εξ αρχής μπορούμε να κάνουμε τις συστάσεις και η αρμοδιότητα αφορά εκείνους οι οποίοι έχουν τα ίνια των δαπανών. Αυτοί πρέπει να ανακτήσουν τα χρήματα. Δεν μπορούμε εμείς να υφαρπάσουμε αυτή την αρμοδιότητα, γιατί έτσι θα τους αποστερήσουμε από το κίνητρο για να δουλέψουν. Αυτό θα ήταν μια απόκληση ούτως υπήρνε από την αποστολή μας. Ε, γι' αυτό και πολλές φορές βέβαια κάνουμε κάποιες συστάσεις που είναι πάρα πολύ απαιτητικέ. ή άλλες φορές, δεν είναι και τόσο σύγχρονο αυτό βέβαια, έχουμε κάποιες συστάσεις όπου βάζουμε τον πύχη πολύ χαμηλά. Άρα χρειάζεται στο σχετικό μέτωπο να δουλέψουμε και άλλο. Για να δούμε τώρα. Με τα δεδομένα που έχουμε όσον αφορά τις ανακτήσεις που έχουμε συστήσει από τη δουλειά μας και με τη βάση των δεδομένων που βρήκαμε, τα κατημέλια θα πρέπει να αναφέρουν σχετικό στην Όλαφ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις συστάσεις επί τη βάση του τι έχουν κάνει. Αυτά από πλευράς δαπάνων σε σχέση με τα διερθωτικά ταμεία και από πλευρά εισοδημάτων. Βλέπετε τώρα το σημείο 14 της έκθεσης τις λεπτομέρειες αυτών των ποσοντρών πλευράς ιδιών πόρων σε σχέση με τις παραδοσιακές ε, ε, εισπράξεις από τους ιδίους πόρους έχουμε δει ότι έχουμε 2,85% 2,58% συγγνώμη από τους ε, συλλεχθέντες ιδίους πόρους αλλά τελικά οι επιπτώσεις ανέχονται το 2,01% δηλαδή αν υπολογίζουμε σωστά οι συστάσεις μας είναι παραπάνω από τις δραστηριότητε ε, ελέγχου ε, των ε, και ερευνών των κράτων μελών. Επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για μια εξαιρετική χρονιά όπου φτάσαμε τα δύο δις ανακτήσεις σε σχέση με την αγγλική περίπτωση, υπόθεση και άλλες υποθέσεις. Αυτά όσον αφορά τους πόρους που Μα έχουν απασχολήσει εμά και τις ε, άλλε αρχέ. Από πλευρά των δαπανών έχουμε συστήσει την ανάκτηση ε, που αντιστοιχεί στο 0,43% του συνόλου των πληρώμων και αυτό αντιστοιχεί στο 1 πέμπτο των επιπτώσεων των συστάσεων των κρατών μελών. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι κακό ω αποτέλεσμα. Για να σα τονίσω όμω τώρα άλλα ζητήματα τα οποία δεν μπορούν να είναι ποσοτικά να αποτιμηθούν αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά για να καταλάβουμε τι κάνουμε για να δούμε πώς τα που θα πρέπει να κινηθούμε στο μέλλον ή να μην κινηθούμε. Πρώτα απ' τα η αποτροπή ε, είναι πολύ σημαντικό το πρόβλημα της αποτροπής μας και αυτό είναι ε, κάτι το οποίο είναι σημαντικό, αλλά δεν μπορούμε να το μετρήσουμε, αλλά δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Επίση το πολυπλασιαστικό αποτέλεσμα, γιατί όταν εστιαζόμαστε σε συγκεκριμένο πρόβλημα ή σε συγκεκριμένο σημείο, έχουμε την αποτροπή, αλλά μπορούμε έτσι να κάνουμε κάποιε αλλαγέ. Και έτσι επηρεάζουμε το γίγνεσθε, ούτω ή στα κράτη-μέλη και στην επιχειρηματική δραστηριότητα των επιχειρηματιών. Τώρα κάνουμε τώρα κάτι διαφορετικό. Για να δούμε πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε κάποια ψηλά στάνταρ επαγγελματικής συμπεριφοράς. Ε, όσον αφορά τα θεσμικά όργανα της εσωτερικής έρευνας, διότι θεώρησα ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι από τη δουλειά μας, κύριε Πρόεδρε, και εσείς ασχολείστε επί πολλά χρόνια με αυτό το ζήτημα. Τι να σας θυμίσω, δεν χρειάζεται για τις έρευνές μας ή για κάποια πραγματικά περιστατικά, τα οποία είναι πολύ επίμαχα. Όλα αυτά για το εσωτερικό των συμβουλών οργανών. Πάντως νομίζω ότι τα πράγματα γνώρισαν μια καμπή, μια αλλαγή τελευταία χρόνια, παρά τα όσα γράφουν τα μέσα ενημέρωσης, τώρα τελευταία. οι πιο δύσκολη τομή είναι τα διευθυντικά ταμεία, ξέρουμε. Και νομίζω ότι έχουμε σημείωση εκεί πρόοδο όσον το τι γίνεται στα θεσμικά όργανα αυτό τον καιρό. Οπότε βλέπετε ότι έχουμε την εντολή ερευνών των μελών, των θεσμικών οργάνων, το προσωπικό σε πολλές περιπτώσεις, σχεδόν σε κάθε περίπτωση. Γιατί έχουμε θέματα απάτης, αμοιβών, επιδομάτων, ιατρικών αποζημιώσεων. Ε, δεν έχουμε κλασικές υποθέσεις και περιπτώσεις διαφθοράς μέσα στα θεσμικά όργανα και να υπάρχει κάποιος συνεργάτης ή κάποιος ειδικός αυτοργός από το εξωτερικό. Έχουμε όμως κάποιες περιπτώσεις. Οπότε έχουμε συνολικά κάνει 17 ε, έρευνες όσον αφορά ε, σοβαρά παραπτώματα στο εσωτερικό των οργάνων. Καταλήξαμε σε 12 συστάσεις και είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το μέτωπο το ότι κάνουμε μία έρευνα. Κάποιος απαλλάσσεται πως έγινε τις τελευταίες μέρες για κάποιον ε, από το Κοινοβούλιο. Διατυπώνονται ισχυρισμοί κατά κάποιου ε, ανωτέρου υπαλλήλου και εμείς θέλουμε να δούμε κατά πόσον συντρέχουν ποινικέ ευθύνε ή εν πάρει περίπτωση Και ακόμα και αν δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε όλα τα στοιχεία, νομίζω ότι πάμε καλά τώρα. Για να δούμε τι γίνεται με τη συνεργασία με τις δικαστικές αρχές. Βλέπετε εδώ ότι και εδώ θα θέξουμε κάτι που συζητήθηκε ήδη σήμερα το πρωί. Ναι, ναι, τελειώνω, τελειώνω πρωί. Σε μία επταετία είχαμε 42% παραπομπές στην δικαιοσύνη σε σχέση με αυτές τις δικαστικές συστάσεις. Βελτιώσαμε τις επιδόσεις μας όσον αφορά τις αποφάσεις κατά τις οποίες δεν ακολουθούν τις τάσεις μας οι εθνικές αρχές και κάθε χρόνο εξετάζουμε κάποια κράτη-μέλη. Το θέμα είναι βέβαια ότι θα μπορούσαν να ασχοληθούν με τις ζημίες βάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ασχολούνται με τη ζημία βάρος του ενό κράτου μέλου, οπότε υπάρχουν στοιχεία ότι δεν ερμηνεύουν κατά τον ίδιο τρόπο όλα τα κράτη-μέλη την κυβερνητική νομοθεσία και άρα κάποια κράτη-μέλη κάνουν παραδεκτά τα στοιχεία που τους δίνουμε πιο εύκολα από άλλα κράτη τα οποία θέλουν να κάνουν τη δική τους έρευνα. Αλλού υπάρχει ταυτόσιμη εθνική νομοθεσία Τσεχία και Σλοβακία μεταξύ τους έχουν ίδια νομοθεσία για προφανείς λόγους. Όμως πάλι η ερμηνεία μπορεί να επικύλει. Και σε άλλα κρατημέλη παρόν. Οπότε και εμείς δεν διστάζουμε να επιληφθούμε κάποιες υπόθεσεις ακόμη και όταν δεν απόκειται σε εμάς να αποφασίσουμε. Θα ήταν λάθος να μην επισημάνουμε ότι υπάρχει θέμα σε κάποια υπόθεση. Και θα πρέπει να δούμε καλύτερα το θέμα των συστάσεων, ακόμα και αν δεν λαμβάνονται υπόψη, να ε, προτάσουμε στις περισσότερες συστάσεις και ας κάνουν ό,τι θέλουν οι υπόλοιποι. Αλλά τέλος πάντων είπαμε ότι οι ρυθμοί ε, ποινικών διώξεων είναι εντάξει σε σχέση και με το παρελθόν. Ελπίζω δεν με ακρηγόρησα, αλλά θέλω να σας πω, αν κατακλείδει, ότι πιστεύω ακράδαντα, όπως λέμε και στην ετήσια έκθεση, ότι παραδίδουμε την σκητάλη ε, με την Όλαφ σε σταθερή ε, ρότα, με την φήμη ότι κάνουμε αντικειμενικά και μερόληπτα τις έρευνές μας και ότι με την καινούργια ηγεσία θα συνεχιστεί στην ίδια σωστή ρότα το, το έργο της ε, Όλαφ Πρόκειται για δουλειά πολλών ανδρών και γυναικών, δεν τους βλέπετε, αλλά θεωρώ ότι είναι τιμή μου να συνεργάζομαι μαζί τους. Και σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Και θα προσπαθήσω στο μέτρο του να τον απαντήσω τυχόν απορίες και ό,τι δεν ξέρω θα το παραπέμψω στο διάδοχο. Ευχαριστώ κύριε Άιλετ και για την εκθεσή σας και το έργο που κρύβεται από πίσω και βεβαίως γιατί τα συγκαρτήριά μου στους συνεργάτες και συνεργάτηδες σας. Έχω μια ερώτηση που θα προτιμούσα να είχα υποβάλει στον ε, προκατοχό σας. Έχω ένα πίνακα, δικός μου είναι ο πίνακας αυτός που δείχνω, με κλεισμένες υποθέσεις και συστάσεις. Γιατί με συστάσεις, διότι αυτές οι υποθέσεις κατέληξαν και σε αποτελέσματα. Σε σύγκριση με τις υπόλοιπες. Για το 2017 βλέπουμε σημαντική μείωση των υποθέσεων οι οποίες βρίσκουν μια συνέχεια. Οι αριθμοί αυτοί προέρχονται από την έκθεση του ίδιου του Όλαφ. Βέβαια θα ήταν ωραίο να μην χρειαζόταν να ψάξω εγώ να βρω τα νούμερα αυτά για να τα βάλω στον πίνακα, αλλά να μας τα είχατε δώσει εσείς. Γιατί δείχνουν την αποτελεσματικότητα και την πραγματική απόδοση της εργασίας του Όλαφ. Είδαμε τώρα η έκθεση περιλαμβάνει πολλές επιμέρους υποθέσεις αλλά δεν υπάρχει μια συνολική επισκόπηση. Διαβάζοντας την έκθεση δεν βλέπω μια συνολική επισκόπηση επί των δραστηριοτήτων και αυτό αποτελεί μια δυναμία της έκθεσης. Οι επιμέρους υποθέσεις βεβαίως είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσε και τις βρίσκουμε καμιά φορά και ε, ε συναρπαστικές και ψυχαγωγικές κλπ. Αλλά προτιμώ μια συνολική επισκόπηση, δηλαδή συγκρισιμότητα με με των αριθμητικών δεδομένων. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Γιατί είναι χαμηλότερα τα νούμερα, ασυνήθιστα χαμηλά σε σύγκριση με προηγούμενα έτη. Έχω πάρει τα νούμερα από το 2002. Είναι εντυπωσιακό λοιπόν, εντυπωσιακή η μείωση αυτή. Δεύτερη ερώτηση. Υπάρχουν δυσκολίες με το σύστημα ηλεκτρονικής επεξεργασίας των δεδομένων. Υπήρξε μάλιστα και ε, απεργία των εργαζομένων το Δεκέμβριο νομίζω. Πού ε, βρίσκεστε το 2016 χρησιμοποίησατε παραπάνω από 50% περισσότερους πόρους για το σύστημα IT και με τις προφορίες που έχουμε εξακολουθεί να μην λειτουργεί το σύστημά σας και πάντως δεν λειτουργεί με τρόπο που να επιτρέπει μια συνολική επισκόπηση για το τι γίνεται και μέσα σε κάθε υπόθεση ξεχωριστά, αλλά και αυτή την επισκόπηση που λέμε, την οποία δεν έχει κανείς διότι το ηλεκτρονικό σας σύστημα είναι πολύ δύσχριστο. Καλά θα ήταν να μπορέσετε να μας πείτε τον σχεδιασμό του Όλαφ για την τροποποίηση του ηλεκτρονικού συστήματος ώστε να σας επιτρέπει απλούστερα να εργάζεστε. Νομίζω ότι γνωρίζετε πολύ καλά γιατί ε, μιλώ. Το τρίτο το περιλαμβάνει η Εποπτική Επιτροπή. Υψηλός αριθμός ανοιχτών θέσεων οργανογράμματος, 6,6%. Δουλειά έχετε όμως αρκετή. Γιατί λοιπόν ε, λείπουν στελέχη. Είδαμε και στα staff reviews όπου ρωτήσαμε δηλαδή ε, συνεργάτες σας μεγάλη δυσαρέσκεια των εργαζομένων στον Όλαφ. Αν μπορείτε να μας πείτε κάτι σχετικά και γι' αυτό. Τι σχεδιάζετε. Έχω και ε, δεκάδες άλλες ερωτήσεις για λεπτομέρειες. Ε, δεν θα τις θέσω τώρα. Θα ήθελα ωστόσο να μπορέσω να τις υποβάλω εγγράφως και να μου δώσετε απαντήσεις. Εξάλλου, σας ευχαριστώ προσωπικά πάρα πολύ για την θαυμάσια συνεργασία τους τελευταίους μήνες. Μπορέσαμε να δούμε και να εξετάσουμε υποθέσεις που απασχολούν τον Όλαφ και μάλιστα είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σε σύγκριση των υποθέσεων του Όλαφ ε, τα τελευταία χρόνια βλέπω μια σημαντική αύξηση της ποιότητας, τουλάχιστον για αυτές όπου μας δώσατε πρόσβαση ε, και γι' αυτό σας ευχαριστώ. Η κυρία Αιάλα Σέντερ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Άιλετ και όλο το προσωπικό της Όλαφ για τα εξαιρετικά αποτελέσματα είναι αλήθεια ότι είναι μια εξαιρετική χρονιά, καθώς ε, η υπόθεση στη Βρετανία σας έδωσε τη δυνατότητα για ανακτήσεις μεγαλών ποσών. Για μας όμως είναι θεμελιώδες να δείξουμε ότι και στην ανάκτηση των κεφαλαίων υπάρχουν εξαιρετικές περιπτώσεις. Και αν δεν υπήρχε η Όλαφ, ε, τότε θα είχαν ε, μείνει στο σκοτάδι τα χρήματα αυτά. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ ε, στο θέμα της εμπειρίας ε, της Όλαφ τελικά. Η πείρα στο ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αυτή που δημιουργεί μία δεξαμενή σοφίας. Και φυσικά λαμβάνουμε την υπόψη και τα λάθη, γιατί χρησιμεύουν ε, ως διδάγματα. Όμως, εγώ θέλω να ρωτήσω από τη σκοπιά των ε, τελωνίων. Μερικές ε, φορές έχουμε τεράστιες ποσότητες φθηνών προϊόντων, όπως είπατε, που βλάπτουν όμως πάρα πολύ τα δημόσια ταμεία και τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά, επ' έχουμε και πολύ πολύπλοκες περιπτώσεις όπου η ανάκτηση των ποσών, ε, ε, μάλλον ότι έχουμε ανάκτηση μικρότερων ποσών, όμως εγώ θέλω να σας ρωτήσω, η ΟΛΑΦ ε, ουσιαστικά πώς παγιώνει ή ε, πώς μέσα από όλα αυτές τις υποθέσεις ουσιαστικά καταλήγει σε ένα θεωρητικό πλαίσιο. Γιατί Κάθε φορά είναι πιο πολύπλοκες ε, οι διαδικασίες, ε, χρειάζονται μεγαλύτερες ε, πληροφορίες. Έτσι λοιπόν αυτή η πείρα της Όλαφ αποτελεί ένα θησαυρό πώς διαρθρώνεται και πώς μπορείτε να βασιστείτε σε αυτή και πώς μπορούμε να βασιστούμε σε αυτή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο. Το 2017 στην έκθεσή σας τονίζονται δύο στοιχεία που νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα και που ξεχωρίζουν ε, σε σχέση με την ε, καθημερινότητα όταν συζητάμε για τα κονδύλια της ε, ΚΑΠ ή των τελωνίων. Πρόκειται για τα κονδύλια για την έρευνα και για την κρίση των προσφύγων. Για τα κονδύλια για την έρευνα, εγώ θα ήθελα να σας συγχαρώ και ε, μπορώ να πω ότι χαίρομαι και πάρα πολύ γιατί είχα μια κάποια αιμονή από μια σειρά input που είχαμε εδώ από διάφορες ε, εκθέσεις που αφορούσαν την γάμα δελτα έρευνας και όταν τελικά κάποιος ε, έβλεπε ε, τα προγράμματα και τα σχέδια τραβούσε τα μαλλιά του. Ε, όμως με ενδιαφέρει πάρα πολύ τώρα να μου δώσετε κάποιες διευκρινήσεις για το πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε ουσιαστικά το θέμα, στην, τα προβλήματα στην έρευνα, γιατί από ό,τι φαίνεται ε, οι επιστήμονες είναι άθικτοι κατά κάποιο τρόπο, δεν μπορούμε να τους θίξουμε. Και ουσιαστικά που πρέπει να δώσουμε την προσοχή ακριβώς σε αυτό το τομέα. Και δεύτερον, έχουμε τα τελευταία χρόνια που υλοποιούμε ε, μία πολιτική απάντησης στην ε, προσφυγική κρίση. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε ακριβώς τι γίνεται με τα τεράστια κονδύλια που επενδύονται για να προετοιμαστεί ένα δίκτυο ασφαλείας της χρήσης αυτών των κονδυλίων. Και επειδή υπάρχει και πίεση από την κοινή γνώμη, συνεχίζουμε να επενδύουμε χωρίς ε, να ξέρουμε πώς ακριβώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε τις διάφορες ε, απόπειρες απάτης. Γιατί ακριβώς ε, αυτοί που εξαπατούν, επαιτεώνες, ουσιαστικά εκμεταλλεύονται μια αδράνεια που μπορεί να υπάρξει. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τη δική σας άποψη σε σχέση με αυτά τα στοιχεία. Ο κύριος Κόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Άιλετ καθώς και τις συνεργάτηδες και τους συνεργάτες σας για την ετήσια έκθεση πεπραγμένων και για την παρουσίαση. Ε, χρειάστηκε να καθίσω στο κάθισμα για να μπορέσω να διαβάσω διότι ζαλίστηκα. Δείχνει όμως και πόσο σημαντική είναι η εργασία σας και πόσο σημαντικά είναι και τα συμπεράσματα που πρέπει να εξαγάγουμε και αν εξετάσω τις απάτες 3,2 δισεκατομμύρια μεταξύ 13 και 16 ή την έκταση των απατών 1,9 ε, ε, δισεκατομμύρια ε, εισαγωγές κινέζικων προϊόντων μέσω Βρετανίας παραποιημένων παπουτσιών και υφασμάτων. Για το θέμα αυτό οργανώνει το γραφείο μου ακρόαση και θέλω να σας ρωτήσω ειδικά για το θέμα αυτό. Πού βλέπετε πρόοδους σε ό,τι αφορά τις καταχρήσεις του τελωνιακού καθεστώτος 42. Πού μπορείτε να διαπιστώσετε κάποιες πρόοδους και πώς βλέπετε την προθυμία των χωρών μελών να συνεργαστούν. Είμαι βέβαιος ότι δεν θα θελήσετε να ονομάσετε χώρες και να πείτε αν συνεργάζονται ή όχι, αλλά πού μπορούμε να ε, ε, βασιστούμε για να πιέσουμε. Ο κύριος Νοβακόφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θυμάμαι πολλές ακροάσεις εδώ στην Επιτροπή μας με προσώπους της Όλαφ. Πιστεύω ότι στο παρελθόν δεν είχαμε τόσους ε, πολλούς λόγους να χαμογελούμε όπως σήμερα. Θυμάμαι, παίρνουμε το ότι για ορισμένε υποθέσει στην αρχή τη εντολή μα, στην αρχή τη θητεία μα, είχαμε τέσσερι ε, φορέ ε, περισσότερε υποθέσει σε σχέση με τι υποθέσει που έκλειναν. Και αυτό ήταν κάπω ύποπτο. Έτσι λοιπόν, καλωσορίζω το γεγονό ότι κλείνουν τώρα οι περισσότερε υποθέσει και υπάρχει και ένα follow-up ε, ω προ τα αποτελέσματα. Όπω βλέπουμε εδώ στο έγγραφο. Επιπρόσθετα, ανησυχώ κάπως για το ότι ένα μέρος της έκθεσης αυτής περιγράφει τις σχέσεις με τα κράτη-μέλη και εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι εθνικές αρχές δεν υιοθετούν τις συστάσεις της Όλαφ, αν και υπάρχουν αποδείξεις είτε ότι έχουν λάβει χώρα απάτες ή λάθη στη χρήση νέων κονδυλίων. Ανοίγει λοιπόν εδώ μία συζήτηση, να βρούμε έναν τρόπο οι συστάσεις της Όλαφ να μην είναι απλώς κάτι στο επίπεδο του ευχολογίου, αλλά να είναι ένα εργαλείο που να πιέσει τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν το κράτος δικαίου όταν υπάρχουν αποδείξεις ε, κακοδιαχείρισης και κατάχρησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Όπως μπορούμε τώρα να κρίνουμε από τα στοιχεία που μας παρουσιάστηκαν. Ε, ο όγκος της δουλειάς της Όλαφ αυξάνεται καθώς ο ευρωπαϊκός προπολογισμός ε, κυρίως ε, σε κάποια κράτη-μέλη φαίνεται να χρηματοδοτεί τις δημόσιες επενδύσεις σε πάνω από 50-60%. Πιστεύετε ότι χρειάζεστε ενίσχυση των ικανοτήτων σας για να μπορείτε να υλοποιείτε περισσότερες έρευνες, να εργάζεστε περισσότερο επιτόπου. Όπως βλέπουμε, αυτό το έργο ουσιαστικά ε, μας προφυλάσσει από κακοδιαχείριση και κατάχρηση δισεκατομμυρίων ευρωπαϊκών κονδυλίων. Έτσι λοιπόν, καθώς ε, τώρα βλέπουμε ότι στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλάσιο υπάρχει μία πρόταση να αυξηθεί ο προπολογισμό πολλών ευρωπαϊκών οργανισμών, ακριβώς γιατί οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε αυξάνονται, ίσως θα μπορούσατε να μπείτε κι εσείς σε αυτή την κατηγορία. Θα ήθελα εδώ να ζητήσω συγγνώμη γιατί μάλλον έχασα αυτό το τμήμα της παρουσίασης αλλά στη σελίδα 4 έχουμε μία αναφορά σε χιλιόγραμμα. Είναι υποθέσεις που συνδέονται με αδήλωτα αγαθά στα τελωνία ή κάτι τέτοιο. Θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις από αυτού λέει εδώ απλώς ποσότητε σε χιλιόγραμμα και υπάρχουν κάποια αριθμητικά στοιχεία που μας δείχνουν διάφορα κράτη-μέλη και τις επιδόσει τους. Σας ευχαριστώ. Thank you. Uh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ξεκινήσω με τις δικές σας παρατηρήσεις για τα στατιστικά στατιστικά στοιχεία, νομίζω ότι πρέπει να δούμε τον πίνακά σα και να δούμε ακριβώ ε, πώ ε, ταιριάζει με το δικό μα. Αλλά θέλω να πω το εξή. Καταρχήν υπήρξαν πολλέ συλλογέ στο πώ εργάζεται η και πώ ε, κάνει διάφορε μετρήσει από το 2002 μέχρι σήμερα. Και είχαμε τουλάχιστον δύο κομβικά σημεία που φαίνεται ότι δεν μπορούν να είναι συγκρίσιμα τα εφημετικά στοιχεία με επιστημονικό τρόπο. Έτσι λοιπόν δεν θα έδινα ιδιαίτερη βάση, πολύ μεγάλο βάρο σε μία απλή παρουσίαση όπως αυτή. Πάντοτε υπήρχε το δίλημα για το να μπορούμε να χρησιμοποιούμε την ίδια στατιστική μέτρηση από χρόνο σε χρόνο που φυσικά βοηθά τη σύγκριση, αλλά μας δυσκολεύει στο να αντικατοπτρίσουμε τον τρόπο που σήμερα λειτουργούμε. Πάντοτε υπήρξε ένα ζήτημα για το πόσο κατάλληλες είναι οι στατιστικές για να εντάσσονται στην ετήσια έκθεση και τελικά δεν χρησιμοποιούμε τόσο πολλά στατιστικά στοιχεία τα τελευταία χρόνια γιατί θεωρήσαμε ότι δεν ήταν ο καλύτερος τρόπος ε, για να επικοινωνήσουμε ευρύτερα όμως γνωρίζω ότι καθιστά πιο δύσκολη την ε, μέτρηση των επιδόσεων. Αν θέλετε βέβαια, θα εξετάσουμε αυτά τα ερευνητικά στοιχεία και θα συζητήσουμε με το δικό σα προσωπικό πώς τα εκεί και θα επανέλθουμε στο θέμα. Η δική μου εντύπωση είναι ότι υπήρχε κάποια μείωση σε κάποια από τα αριθμητικά στοιχεία το 2017 για διάφορους λόγους, ε, το σύστημα πληροφορικής, το οποίο θα αναφερθώ σε λίγο αλλά και επειδή ιδιαίτερε προσπάθειε έγιναν τα προηγούμενα έτη να ξεκαθαρίσουν οι παλιές υποθέσεις. Και πετύχαμε και ένα μερικό αποτέλεσμα. Είχαμε πολύ δεχτερή μείωση ε, την ε, στιγμή που αναλαμβάνουμε τις έρευνες. Έτσι λοιπόν ε, θα ήμουν κάπως προσεκτικός στο να προωθήσω, να το σπρώξω αυτό παραπέρα γιατί αν περιορίσουμε και άλλο το χρόνο των ερευνών, θα έχουμε και πλήγμα στην ποιότητα. Σε ό,τι αφορά τώρα τα συστήματα πληροφορικής, ε, το οποίο λέγεται το σύστημα αυτό OCM, υπάρχουν δυσκολίε. Έχουμε αντιμετωπίσει πιο πολλέ δυσκολίε από ό,τι περιμέναμε. Πέρσι, τι κάναμε. Επανήλθαμε στα βασικά και ουσιαστικά διορθώσαμε κάποια στοιχεία στην καρδιά του συστήματος, στις βασικές λειτουργίες, έτσι ώστε να λειτουργεί καλύτερα. Είχαμε και επιπλέον εμπειρογνώμονες που μας έδωσαν συμβουλές για το ότι δεν πήγαινε καλά. Τώρα, έχουμε με ηλεκτρονική ε, ροή εργασίας που δεν είχαμε στο παρελθόν. Στο παρελθόν είχαμε σωρούς από χαρτιά που τα κουβαλούσαμε γύρω-γύρω στα κτίρια από διάφορους ανθρώπους, γραμματείς κτλ. Όσο αυτό έχει σταματήσει τώρα και είναι πραγματική βελτίωση της ασφάλειας. Είναι καλύτερη κατάσταση. Δεν σας κρύβω ότι εξακολουθούμε να έχουμε προβλήματα. Όπως και πολλοί άλλοι που είχαν ιδιαίτερα φιλόδοξα προγράμματα και ίσως θα χρειαστούν ακόμη 2-3 χρόνια από αυτό που ελπίζαμε πριν έχουμε την ε, λειτουργία στο 100%. Βέβαια, οι βασικές ε, λειτουργίες ε, υλοποιούνται σήμερα καλύτερα και γρηγορότερα και πολύ προσεκτικά. Σιγά σιγά θα έχουμε νέες λειτουργίες. Και επίσης θα πάρουμε λίγο περισσότερα χρήματα για να προσπαθήσουμε να προσλάβουμε τους σωστούς ανθρώπους ε, δυνάμει και των διαθέσιμων κονδυλίων για να κάνουν τη δουλειά. Αλλά έχουμε ανθρώπους που είναι ιδιαίτερα φασιωμένοι να το διορθώσουν αυτό, να το κάνουν σωστά και νομίζω ότι με κάποια πίεση θα φτάσουμε τελικά στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμη όμως. Υπάρχει κάποιος ε, αξιόλογος αντίκτυπος δηλαδή κυρίως ό,τι αφορά τις ε, αξιολογήσεις, γιατί οι πρώτοι που ήταν ε, στην πρώτη γραμμή ήταν ε, οι άνθρωποι οι οποίοι συνέστηναν ότι θα έπρεπε να ανοίξει όχι μία έρευνα. Και έχει επιβραδυνθεί η δουλειά σε μεγάλο βαθμό λόγω των δυσκολιών που είχαμε με το σύστημα. Αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση παρά να συνεχίσουμε με αυτά που κάνουμε δεν μπορούμε να σταματήσουμε και να κάνουμε κάτι άλλο, θα πρέπει να λειτουργήσει. Και αυτό θα κάνουμε. Σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις στο προσωπικό, ούτε και εμείς είμαστε ικανοποιημένοι μας διαβάσαμε, που έχει να κάνει και με κάποια γεγονότα του παρελθόντος. Θα κάνουμε μια έρευνα δεν γίνονται αυτέ οι έρευνε κάθε χρόνο, αλλά θα κάνουμε μια έρευνα να δούμε τι πιστεύουν τώρα οι άνθρωποι και ίσως να έχουν αλλάξει οι συνθήκε τον τελευταίο καιρό. Θυμάμαι ότι είχαμε έναν προηγούμενο πρόεδρο τη Εποπτική Επιτροπής, ο οποίο με τη μακρά πείρα του έλεγε ότι τείνουμε να πετυχαίνουμε χαμηλότερα αποτελέσματα από φορείς ε, που η εργασία τους δεν ενοχλεί τόσο τις κυβερνήσεις. Βέβαια, έχουμε μια ολόκληρη στρατηγική για να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Από την καλύτερη επικοινωνία μέχρι δραστηριότητες, την ε, building. Μάλιστα, είχαμε και σε έναν αγώνα μπάσκετ, έκανα και έναν αγώνα μπάσκετ ε, πριν κάποιες εβδομάδε. Ε, να αναγνωρίσουμε βέβαια ότι είναι ένα θέμα στο οποίο πρέπει να εργαστούμε περιττέρω. Αν μπορώ να περάσω τώρα στα σχόλια της κυρίας Αγιάλα Σέντερ. Και εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένο για τα όσα συνέβησαν στον τελωνιακό τομέα. Έχουμε διάφορα είδη εμπειρογνωμοσύνη. το χάρη, έχουμε ανθρώπου που είναι πολύ εξοικειωμένοι με την αγορά τη επί επιτόπου. και πολλές επιχειρησιακές αποστολές ε, στις χώρες όπου παράγονται αυτά τα προϊόντα. Υποτίθεται ότι παράγονται. Αλλά έχουμε και εμπειρογνώμονες ε, στα λογιστικά. Η περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου αφορούσε πολλά δεδομένα και οι εμπειρογνώμονες στον τομέα αυτό έχουν αποκτήσει τώρα μεγάλη φήμη, όχι μόνο στις ευρωπαϊκές τηλεονικές υπηρεσίες, αλλά και στην Κίνα και αλλού. Για το φως που μπόρεσαν να ρίξουν στην υπόθεση και την ταχύτητα με την οποία αντέδρασαν. Και έχουμε εμπειρογνώμονες και σε άλλους τομές, όπως οι προδρομές ουσίες, και φυσικά και για τα τσιγάρα παραδοσιακά, αλλά και σε άλλους μυς, παίρνουν το σχάρι, τα ποδήλατα, το fasteners, πώς το λέμε, θυμάμαι. Όμως, οι τελωνιακοί δασμοί είναι πηγή εσόδων. Έτσι λοιπόν είναι το παραπροϊόν της βιομηχανικής πολιτικής. Που έχει να κάνει και με τους ε, δασμούς αντι-dumping. Τα κράτη-μέλη συνηθίζουν να θεωρούν τους τελωνιακούς δασμούς δεδομένους και να θέτουν πόρους αλλού. Να σχολιάσω εδώ κάτι που υπόθηκε ότι πολλά από αυτά τα θέματα σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα των πόρων στα κράτη-μέλη και με την κατανομή των πόρων. Αν και τώρα πάει δεν πειράζει, γιατί τα κράτη-μέλη τείνουν να επικεντρώνονται, παραδείγματο χάρη στι απάτες με τον καπνό ή στην ε, θέμα τη ασφάλειας ή και στα δύο. Αλλά φυσικά θα υπάρχουν ε, επιπτώσεις για τη δουλειά τη συλλογή εισόδων πρέπει να γίνει από την ίδια υπηρεσία. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα έχουμε υπό εξέταση και ξέρω ότι η ΓΔ στην ΓΔ ΤΑΞ και budget φτάζουν αυτά τα θέματα με ναι, προσοχή, με ενωμένη προσοχή είπα το φως της δουλειάς που κάνουμε. Τώρα για τις δαπάνες ε, για την έρευνα. Είναι πολύ σαφές τι προβλήματα έχουμε. Συχνά δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, αλλά είναι δύσκολο σε ένα συγκεκριμένο τομέα να αντιδράσουμε. Πολλές φορές ε, υπάρχει ένα τέλος ε, για το ίδιο έργο ή μπορεί το χάρη να ισχύει για κάποιο τύπου είναι σκουπίδι και στις ορισμένες περιπτώσεις είχαμε προγράμματα όπου η απέτηση είναι ο να διαμένει σε ένα συγκεκριμένο μέρος προκειμένου να οικοδομήσει, να χτίσει μια δουλειά μεταξύ των πανεπιστημίων και να δώσει στους ανθρώπους ε, το μήνυμα για το τι σημαίνει Ευρώπη. Αλλά φυσικά με το διαδίκτυο δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό για να κάνεις την έρευνα. Δεν ακολουθούν όλοι τους ε, κανόνες ε, και εκεί είναι κάπως τίθεται το θέμα πώς θα πάρουμε πίσω τα χρήματα. Τώρα για τους πρόσφυγες. Βεβαίως. Όλοι ασχολούνται με αυτό, κυρίως όσοι είναι υπεύθυνοι για τις δαπάνες, γνωρίζουν τους ε, κινδύνους που ενέχονται στην ε, παράδοση έκτακτης βοήθειας σε επικίνδυνα μέρη και έχουν συστήματα, ενώ φυσικά να γνωρίζουν ότι υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να γίνει στην επιβολή και πρέπει να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ της εξοικονόμησης πόρων και της διάσωσης ζώων. Έτσι λοιπόν τα γνωρίζουν όλα αυτά και εμείς συνεργαζόμαστε μαζί τους και τους δίνουμε συμβουλές και μας τηρούν ενήμερους. Όμως ο κίνδυνος βεβαίως είναι ότι θα πούνε οι άνθρωποι ότι υπάρχουν οι κίνδυνοι αυτοί Επομένως είναι απαραίτητο να δαπανώνται χρήματα με ένα ταχύ σύστημα ε, δημοσίων συμβάσεων, γιατί είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα, ενώ μπορεί να μην είναι και τόσο. Και φυσικά εκεί πρέπει να δίνουμε πολύ μεγάλη προσοχή και έχουμε μια σειρά ερευνών, όπου ο ισχυρισμός, μάλλον όπου εμείς ε, δοκιμάζουμε την υπόθεση ότι οι μηχανισμοί ε, παροχής έκτακτης βοήθειας ε, δεν ήταν απαραίτητη. Προσπαθούμε να εκπονήσουμε μία έκθεση όπου τουλάχιστον όσοι είναι υπεύθυνοι για την ε, δαπάνη των χρημάτων να μπορούν ουσιαστικά να διωχθούν ή να τους επιβληθούν κάποιε κυρώσει ε, αν ε, πρόκειται σε Για να πάω τώρα στα σχολεία του κ. Νόβακου. Γιατί δεν θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση στα κρατημέλη για follow-up. Σίγουρα δεν έχουμε νομική βάση να το κάνουμε αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι θέμα αρχής γιατί οι αποφάσει περί ανάκτηση κονδυλίων και το πόσο κονδυλία θα ανακτηθούν θα πρέπει να λαμβάνονται από αυτού που έχουν δαπανίσει τα χρήματα υπό το φω των πληροφοριών που του δίνουμε και θα πρέπει να λογοδοτούν. Δέχομαι ότι μπορούν και τέλειοι ηλεκτρικοί μηχανισμοί, οι μηχανισμοί λογοδοσία, όμω είπατε, κύριε Πρόεδρε, ότι η Επιτροπή σα έχει ένα πολύ ισχυρό μηχανισμό λογοδοσία. Υπάρχουν και άλλοι στα κράτη-μέλη που κάνουν την ίδια δουλειά. Βεβαίω και δεν θέλαμε περισσότερε πληροφορίε. Όταν δεν μα λένε γιατί δεν έχουν υιοθετήσει τι συστάσει μα και θέλουμε ισχυρότερου μηχανισμού, τουλάχιστον αυτοί που δεν του ακολουθούν να μα εξηγήσουν γιατί δεν το κάνουν. Τώρα, οι περαιτέρω ικανότητε ε, σε σχέση με το διαφορετικό ταμείο είναι ένα θέμα. Κύριο Κέσλερ ενδυνάμωσα το input που έχουμε βάλει στα διευθυντικά ταμεία. Εμεί ε, μετακινήσαμε για κάποιους ανθρώπους σε αυτές τις μονάδες και τώρα κατόπιν διαγωνισμού μπορούμε να προσλάβουμε περισσότερους ερευνητές ε, με ειδικέ γνώσεις ε, όμως ε, πρέπει να εργαστούμε στις γλώσσες του κράτους μέλους. Μπορεί να τους χάρη να μην έχουμε ανθρώπους που να μιλούν μια συγκεκριμένη γλώσσα και μπορεί να υπάρχει ένα εμπόδιο εκεί. Και αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν θα ξεκινήσουμε μία έρευνα, δεν θα ανοίξουμε μία έρευνα στη χώρα τάδε, γιατί δεν έχουμε διαθέσιμους ερευνητές. Ενώ αν τα ίδια γεγονότα συνδέονται με την μία άλλη χώρα, την Υψηλόν, μπορεί να είχα τους κατάλληλου ερευνητέ. Δεν είναι ιδανική κατάσταση, αλλά έτσι είναι. Και φυσικά χάσαμε και τις πόρους, για λόγους που όλοι κατανοούμε. Τώρα έχει σταματήσει αυτό. Ένα κύριο ζήτημα είναι αν η δουλειά της Άλαφ θα είναι ουσιαστικά χρήσιμη από το παρόντος όταν θα ξεκινήσει και το έργο της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Συγκυρία σε λίγα χρόνια. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα αυξηθεί η δουλειά για την όλα. Με την ΕΠΟ παρά θα μειωθεί. Θα πρέπει να σκεφτούμε βέβαια και δημοσιονομικά θέματα με αυτό το χρόνο και ο διαδοχός μου μάλλον θα ξοδέψει ένα μεγάλο μέρος της θητείας του για να σκέφτεται αυτών των πραγμάτων. Όμως αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι πραγματικά πράττουμε τα όσα πρέπει σε ό,τι αφορά τις έρευνες στα διαφορετικά ταμεία, ε, στα κράτη-μέλη, όπου υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα. Κάποια είναι παλιά κράτη-μέλη, κάποια άλλα όχι. Νομίζω όλοι ξέρουμε σε τι αναφέρομαι. Και έγινε και μια αναφορά στα εγκλωστευοντουργικά Κοιτάξτε, όταν είναι φθηνά τα κλειστοφωτιουργικά, τα μετράμε με το βάρος παρά με τον αριθμό ε, των ε, τεμαχίων. Για να σας απαντήσω. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ να απαντήσω στις ερωτήσεις. Η Πρόεδρος κυρία Γκρέσλε, ευχαριστώ πολύ. Επισημένω, διότι είπατε ότι θα ήταν πιο απλό. Τα νούμερα αυτά τα έχω πάρει από τις αιτήσεις εκθέσεις του Όλαφ και είναι οι ε, υποθέσεις που έχουν κλείσει με follow-up. Βρίσκεται και τις ε, total closed cases εδώ. Δεν βλέπουμε όμως πια το συνολικό αριθμό των κλειστών υποθέσεων. Ε, προκύπτει μόνο από τον πίνακα που έχω συντάξει εγώ η ίδια. Δεν βλέπουμε επίσης πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την διάρκεια των ερευνών έχω την εντύπωση ότι όταν βολεύει εμφανίζεται το στοιχείο αυτό, όταν δεν βολεύει δεν εμφανίζεται. Μα λείπουν κάποια λοιπόν βασικά δεδομένα. Ορίστε κύριε Άιλετ πάλι αν θέλετε να απαντήσετε. Κύριε Πρόεδρε, σελίδα 53 του στατιστικού παραρτήματος εκθέσεω. Μου φαίνεται ότι περιλαμβάνει πολλές πληροφορίες σχετικά με αυτά τα πράγματα που ε, λέτε. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν θα θέλατε η συνεδρίαση να γίνει στατιστικό σεμινάριο, αλλά ε, περιλαμβάνουμε πολλές σχετικές πληροφορίες στο παράρτημα που σας είπα, η Πρόεδρος. Μέχρι τώρα, ε, investigations concluded ήταν κάτι διαφορετικό από investigations closed. Γι' αυτό πήραμε τα νούμερα για τις investigations closed. Πρόκειται για θέμα ορολογίας, το οποίο θα το θέσουμε και πάλι βέβαια. Ρωτώ σχετικά με το ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο είναι βέβαια βασικό εργαλείο για την δουλειά του Όλαφ. Πώς βλέπετε τα επόμενα βήματά σας, δηλαδή τι πρέπει να γίνει ώστε το ηλεκτρονικό σας σύστημα είναι πραγματικά αξιόπιστο και αποτελεσματικό και να μπορείτε πραγματικά να δουλέψετε ως ερευνητής του Όλαφ, ως ε, χρήστης που ε, καλείται να το χρησιμοποιήσει. Σας παρακαλώ λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, έρευνα που έκλεισε και ολοκληρώθηκε είναι συνώνυμα για μας. Δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτή η παρέξη τώρα όσον αφορά το σύστημα της ε, πληροφορικής. Εν μέρη. το θέμα είναι πώς θα είναι ταχύτερο παρά τους μηχανισμούς ασφαλείας, τις ασφαλιστικές λικλίδες, η καταγραφή κάθε πατήματος κουμπιού που είναι περίπου των τέταρτων των δεδομένων που σώζουμε όσο πιο πολύ ασφάλεια τόσο το σύστημα γίνεται πιο αργό και φυσικά ενοχλητικό πρέπει να περιμένει κανείς. Α, και για, το, για τα έγγραφα σε χαρτί περιμέναμε. Κι εγώ δουλεύω σε δύο ταυτόχρονα υπολογιστές. περιμένω ο ένας να κάνει τη δουλειά του και ε, πρέπει να περιμένω 20 έγγραφα να βγουν να υπογραφούν και εγώ εντωμεταξύ στέλνω κάποια mail, τι να κάνουμε. Δεν μπορεί να είναι τέλεια. Ε, πρέπει να δουλεύουμε με ρυθμούς που επιβάλλουν οι μηχανές και πρέπει να έχουμε το λογισμικό το οποίο πρέπει να το υποστηρίζουν οι τεχνικοί. Τώρα, οι μηχανές αναζήτησης επίσης πρέπει να δουλεύουν πιο γρήγορα για να μπορούμε να αντλήσουμε από το σύστημα τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Για την διαχείριση των πραγμάτων. Και έχουμε αυτούς τους ερευνητέ οι οποίοι πρέπει να μπουν στο σύστημα. Πολύ σημαντική δουλειά τους. Το έργο τους είναι πολύ ικανοποιητικό. Αλλά έχουμε και κάποιους εξειδικευμένους τομείς όπου πρέπει να δουλέψουμε με ηλεκτρονικό ταχυδρόμιο. Και μην πρέπει να καλύψει τα πάντα το σύστημα πληροφορικής που υπάρχει. Ε, είναι, είναι φιλόδοξες προσδοκίες σε αυτό το μέτωπο. Ήδη έχουμε πετύχει πολλά, αλλά όπως γίνεται πολλές φορές με νέες προσπάθειες, δεν μπορεί να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Και βέβαια και θέμα επικοινωνίας του προσωπικού. Γιατί αυτό που στον κοινό χρήστη φαίνεται μια απλούστευση όταν κανείς μιλάει με αυτούς που κάνουν το πρόγραμμα τότε αυτοί το θεωρούν απλούστευση το αυτό που ζητάμε το θεωρούν ε, μπέρδεμα, περίπλοκο οπότε πάντα υπάρχει αυτή η προστριβή μεταξύ χρηστών και προγραμματιστών Δύσκολο να σας πω ακριβώς τι χρειαζόμαστε των προτέρων και να κάνουμε την παραγγελία. Οπότε μόνοι μας φτιάξαμε το σύστημα και αυτό ήταν δύσκολο στο ιστορικό της υπηρεσίας. Τα καταφέραμε και νομίζω ότι θα τα ξανακαταφέρουμε. Το δε κόστος λειτουργίας εάν δεν χρειάζεται βελτίωση, είναι περίπου μισό εκατομμύριο εκατομμύριο, δισεκατομμύρια. 500.000 ευρώ ετησίως. Ε, έχουμε τη βελτίωση, πάμε στο 1,2 εκατομμύρια ετησίως για 2-3 χρόνια ακόμα. Σας ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις. Ήρθαμε στο τέλος τώρα της ε, ε, υποθέσεως αυτής, δηλαδή του θέματος αυτού. Θα μείνετε νομίζω, έτσι δεν είναι. Να δώσω το λόγο στον κύριο Γιάν Μούλντερ, πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας του Όλαφ, για το επόμενο θέμα, ε, θέμα ε, της δραστηριοτήτων Επιτροπής Εποπτείας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας κατά πολέμηση της απάτης. Θα κάνω μια μικρή εισαγωγή και κατόπιν ο συνάδελφος θα πάρει το λόγο. Καταρχήν, ε, ο χρόνος που πέρασε ήταν για την Επιτροπή Εποπτείας μια μεταβατική περίοδος. Όλα τα μέλη σχεδόν είναι καινούργια. παρατήθηκε ο Γενικός Διευθυντής και έπρεπε να ε, μεταφέρουμε τη γραμματεία από την Όλαφ ε, στην ΠΜΟ και φυσικά υπήρξε μια αναταραχή. Αν διαβάσουμε τις προηγούμενες αιτήσεις εκθέσεις, τονιζόταν ότι η Επιτροπή ένιωθε ότι δεν μπορούσε να λειτουργήσει γιατί δεν είχε πρόσβαση στις ε, πληροφορίες που επιθυμούσε. Η Επιτροπή έπρεπε να αποπτεύει την Όλαφ, αλλά ήταν στη διακριτική ευκαιρία της Όλαφ να παρέχει τις πληροφορίες ε, που θεωρούσε απαραίτητες για να ελοπίσουμε εμείς το δικό μας καθήκον. Από την αρχή είπαμε ότι η κατάσταση αυτή δεν είναι αποδεκτή και θα αναφέρουμε τώρα με ικανοποίηση ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση σημαντικά. Τώρα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Άιλετ, ο οποίος έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στην παροχή των πληροφοριών. Ήταν παρόν ε, σε όλες ε, σχεδόν τις συνεδριάσεις που είχαμε, μας έδινε τις κατάλληλες πληροφορίες και εμείς θεωρήσαμε ότι αυτό ήταν πολύ σημαντικό. στον κύριο όγκο της εργασία μας είχαμε την, Excel, την αξιολόγηση του κανονισμού 883, το συζητήσατε σήμερα το πρωί. Υλοποίησαμε μια σειρά συστάσεων. Ορισμένες αντικατοπτρίζονται στην πρόταση της Κομισιόν, ενώ άλλες όχι. Το Σεπτέμβριο ίσως μπορούμε να σας στείλουμε κάποιες άλλες συστάσεις που θεωρούμε ότι λείπουν από την οδηγία. Όμως τα κύρια σημεία είναι το εξή πρέπει να τονίσουμε ότι η Επιτροπή έχει δικαίωμα στην ενημέρωση. Δεν είναι κάτι εξειδικευμένο. Θέλουμε μεγαλύτερη σαφήνεια για τις δικονομικές εγγύησεις και αναφέρθηκε και στη συζήτηση. Επιθυμούμε η συνεργασία των κρατών μελών με την Όλαφ να γίνει υποχρεωτική. Η διαδικασία προσλήψεων για τον νέο Γενικό Διευθυντή ήταν αντικείμενο παρατήρηση από την Επιτροπή μας σε όλα τα στάδια. Εμείς θέλουμε να βελτιώσουμε τη διαδικασία και μπορούσαμε να το πράξουμε. Όπως πάντα, θεωρούσαμε ότι είναι δυνατόν κάποιες βελτιώσεις να γίνουν όμως γενικά θεωρήσαμε ότι μπορούμε να δώσουμε θετική ετοιμαγορία για όλη την διαδικασία πρόσληψης. Και ε, μπορεί ο κύριος Κέσλερ να διοριστεί. Στην έκθεσή μας επίσης αναφέρουμε κάποια κρεμή ζητήματα. Θέλουμε του χρόνου να επικεντρωθούμε και δεν ξέρω πότε, αλλά νομίζω ότι στην επόμενη της έκθεσή μας θα αναφερθούμε περισσότερο. Αλλά θα θέλαμε να τηλοποιήσουμε τις δικονομικές εγγύησεις. Πιστεύουμε αυτή τη στιγμή ότι δεν είναι επαρκώς ικανοποιητικό το σύστημα. Ιδίως η διαδικασία καταγγελιών θα μπορούσε να βελτιωθεί. Όμως θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα μόνιμο σύστημα, έτσι ώστε να μπορούμε να εγγυηθούμε καλύτερα αυτά που απαιτούνται στον κρονισμό. Θα ήθελα να επικεντρωθώ και στη διάρκεια των ερευνών και θέλουμε και να επικεντρωθούμε σε όσο τονίστηκα στη συζήτηση να βελτιώσουμε τα ποσοστά επιτυχίας με τις εθνικές αρχές. Αυτά είναι τα κυρία σημεία, Πρόεδρε. Εισαγωγικά από μένα. Και αν μου επιτρέπετε, ήθελα να δώσω το λόγο στην Ελένα Φασέντα, η οποία θα μας παρουσιάσει μια σειρά άλλων τυχών της έκθεσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Ε, σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα να παρευρίσκομαι εδώ. Και όπως τονίσαμε, η Επιτροπή Εποπτείας γνωρίζει ότι η κύρια προτεραιότητά της ε, ήταν κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής ε, περίοδου ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε η ενίσχυση της ανεξαρτησίας ε, της ερευνητικής δραστηριότητας της Όλαφ. Και γι' αυτό είναι απαραίτητο η Επιτροπή αυτή, όπως είπε και ο Πρόεδρος, να διαθέτει κάθε πληροφορία και επίσης ε, τα υλικού και τους ανθρώπινους πόρους ε, που είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση της αποστολή της. Στο πλαίσιο αυτό θα θέλαμε να εκφράσουμε τη δυσαρεσκιά μας, όπως αναφέραμε και στην έκθεσή μας, ότι η κατάσταση της γραμματείας ε, και οι αλλαγές δεν ανταποκρίνονται στις αναγκαιότητες της γραμματείας, ούτε της Επιτροπής. Όμως, όταν ε, έχουμε κατά νου την ανεξαρτησία, πώς πρέπει να δράσουμε εμείς ως Επιτροπή για να την ενισχύσουμε. Έχουμε κάποια σημεία που έχουμε ήδη εντοπίσει ως πρωταρχικά. Καταρχήν, μέσω του τακτικού ελέγχου των ερευνών της Όλαφ. Πράγματι, ο πραγματικός έλεγχος είναι το κύριο εργαλείο που διαθέτουμε διαθέτει η Επιτροπή μας για να διασφαλίσουμε ότι δεν έχουμε εξωτερικές παρεμβάσεις ε, στην άσκηση ε, της ε, λειτουργίας της έρευνας και των να υιοθετούνται οι δικονομικές αποφάσεις σύμφωνα με τις αρχές νομιμότητας, αμεροληψίας και του απόλυτου σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των δικονομικών εγγύσεων. Δεύτερον, επίσης όπως τονίσαμε στην γνωμοδότησή μας 2-2017, κατανοούμε ότι τα διαρθρωτικά προβλήματα που αναφέρουμε εκεί, παραδείγματο χάρη η εσωτερική οργάνωση της Όλαφ, αποτελούν ε, έναν ε, ενδυνάμει κίνδυνο για την άσκηση της ανεξαρτησίας των ερευνών. Τρίτον, αναφερόμαστε στην ε, ενίσχυση της ανεξαρτησίας. Είναι κάτι απολύτως απαραίτητο, όχι μόνο τη στιγμή της απόφασης για το αν θα ανοίξει ή αν δεν θα ανοίξει μια έρευνα, αλλά επίσης ε, και στις ε, δύο συγκεκριμένες δικονομικές στιγμές που ακολουθούν, δηλαδή την υλοποίηση της έρευνας και τη στιγμή που κλείνει η έρευνα ως προς τη στιγμή της ε, λήψης της απόφασης για το αν θα ανοίξει μια έρευνα ή όχι, η Γραμματεία και αυτή η Επιτροπή με την υποστήριξη της Γραμματείας αναλύει τις ε, πληροφορίες ε, που έχουν ληφθεί από την Όλαφ σε σχέση με τις 60 dismissed cases, δηλαδή πληροφορίες που έλαβε η Όλαφ από διάφορες πηγές από ιδιώτες ε, ή από την Κοινωνική Επιτροπή ή πληροφορίες που λάβαμε από άλλους ευρωπαϊκούς ε, φορείς και αποφάσισε να μην ανοίξει έρευνα για τις υποθέσεις αυτές. Πέμπτον, τονίζουμε σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα στην ε, υλοποίηση και την ανάπτυξη της έρευνας, τονίζουμε ότι η Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε συγκεκριμένα σημεία που είναι τα εξής, η διάρκεια των ερευνών και ο σεβασμός για τις προθεσμίες της έρευνας που θα πρέπει να υλοποιείται χωρίς διακοπή κατά τη διάρκεια μιας περίοδου που θα πρέπει να είναι ανάλογη σε σχέση με τις συνθήκες και την πολυπλοκότητα της υπόθεσης για να αποφύγουμε την παραγραφή των ε, ερευνών όπως ε, θα αναφερθεί και στη συνέχεια από τη συνάδελφο. Λοιπόν, ε, σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικονομικών εγγυήσεων που είναι η συγκεκριμένη έκφραση της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας της Όλαφ στην εκτέλεση των ε, εξουσιών έρευνα και συγκεκριμένα το δικαίωμα των διαφερωμάτων να εκφραστούν επί των γεγονότων και επίσης αυτό αποτελεί μια κυρία ανησυχία στο έργο της Επιτροπής. Μια άλλη πολύ ευαίσθητη στιγμή έχει να κάνει με το εξή. Ε, έχει να κάνει με τη στιγμή που ξεκινάει η έρευνα και τη στιγμή που κλείνει συγγνώμη, η έρευνα και, με το αν θα εκπονηθούν ε, ή όχι συστάσεις από το Γενικό Γραμματέα της Όλαφ. Η μόνιμη πρόσβαση της Επιτροπής επομένως στις πληροφορίες μέσω μιας μόνιμης δομής, ε, όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος, είναι θεμελιώδης για την Επιτροπή προκειμένου να μπορέσει να βοηθήσει το Γενικό Γραμματέα το Γενικό Διευθυντή, συγγνώμη, στην ε, υλοποίηση των καθηκόντων του και να εγγυηθεί την ανεξαρτησία του. Η Επιτροπή αυτή, για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, αυτή τη στιγμή εξετάζει τέσσερις έρευνες που έχουν ολοκληρωθεί, μία με συστάσεις και άλλες χωρίς συστάσεις. Με ξεκάθαρο τρόπο θέλουμε να πούμε ότι οι γνωμοδοτήσεις για τα θέματα αυτά αποτελούν ε, προτεραιότητα στο σχέδιο εργασίας ε, της Επιτροπής αυτής για το τρέχον έτος 2018. Όμως, ε, στην πραγματικότητα, οι δυσκολίες που έχουν εντοπιστεί σε επίπεδο γραμματείας βεβαίως και θέτουν κάποια θέματα που αφορούν την ολοκλήρωση των εργασιών. Όμως αυτή, αυτό το έργο αποτελεί πράγματι προτεραιότητα για το 2018. Θα ήθελα τώρα να αναφέρω μία άλλη πτυχή που έχει να κάνει με τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, της ΕΠΟ και της ΕΟΛΑΦ. Και πιστεύω ότι όλοι γνωρίζουμε ότι η ΕΟΛΑΦ ε, ήταν και θα συνεχίσει να είναι Ιδίω στα κράτη-μέλη που δεν έχουν προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο μόνος ευρωπαϊκός οργανισμός που εξειδικεύεται στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωση η Επιτροπή, με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ε, και ε, γνωρίζει και την ε, απόφαση του Ευρωπαϊκού το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Μαΐου 2018 έλαβε λοιπόν υπόψη την έκθεση για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η Επιτροπή ε, προσδιορίζει ως ε, ένα από τα κύρια καθήκοντά του στο εγγύς μέλλον το να συνεισφέρει ενεργά για την οικοδόμηση των σχέσεων μεταξύ Όλαφ και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Με την έννοια αυτή, η Επιτροπή ήδη εξέφρασε ότι η μελλοντική επιχειρησιακή σχέση μεταξύ της όλαφε και της εισαγγελία είναι μια ευκαιρία για την όλαφε να εξυγχρονίσει την ε, λειτουργική και οργανωτική δομή της αλλά και τις αρμοδιότητές της στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του κανονισμού όπως υπόθηκε και σήμερα το πρωί η Όλαφ είπε ότι πρέπει να δώσει υψηλού επίπεδου αρρωγή στην Ευρωπαϊκή Συγκυλία και ότι όπως λέει και το Κοινοβούλιο στον λογοψήφισμα και στο πλαίσιο της αναθεώρησης του κανονισμού 883 του 2013 και παραθέτω να δημιουργήσει μια κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των αρποδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Αγγελία και της Όλαφ προκειμένου να ενισχύσει τις δικονομικές εγγύησεις, να ξεκαθαρίσει και να ενισχύσει τις ε, αρμοδιότητες έρευνας της Όλαφ και να δημιουργήσει ένα επίπεδο διαφάνειας σε σχέση με τις συστάσεις ε, και τον ε, εκθέσεων της Όλαφ και να ξεκαθαρίσει τους κανόνες σε σχέση με τα δεδομένα συνεργασίας μεταξύ Όλαφ και της Επιτροπής Ελέγχου. Η σχέση μεταξύ Όλαφ και Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν θα υλοποιηθεί από τη μία μία μέρα στην άλλη. Και φυσικά το γνωρίζουμε αυτό. Αντιθέτως, εμπειρία που έχουμε Δηλαδή με την έννοια της συνεργασία με τον, μεταξύ των δύο, πέρα από ξεκαθάρισμα του κανονισμού, θα χρειαστεί ένα μεγάλο αριθμό λύσεων που πιθανότητα θα περάσουν από συμφωνίες, πρωτόκολλα, από νέες καταστάσεις, αμφίβολες, που όλες θα πρέπει να ξεπεραστούν χρησιμοποιώντας τη γνώση μας, την εμπειρία μας και ε, την εξειδίκευση όλων των ενδιαφερομένων, των εχομένων Και σε αυτό ακριβώ το πλαίσιο η Επιτροπή Εποπτεία ε, με την 20η πείρα τη ε, είναι διατεθειμένη να συνεισφέρει για μια επιτυχή σχέση μεταξύ Όλαφ και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα, ένα άλλο σημείο που θα ήθελα να θίξω σχετίζεται άμεσα με τις προτεραιότητες της πολιτικής έρευνας. Η Επιτροπή επίσης ε, έχει λάβει υπόψη την ανακοίνωση ε, του Προέδρου ε, της Επιτροπής, της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027. Εδώ εξηγείται η πολιτική των δημοσιονομικών προτεραιοτήτων. Η Επιτροπή διεξέφρασε την άποψή της στην ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ε, διάφορων θεσμικών οργάνων τον περασμένο Νοέμβρη και υιοθετεί εκ νέου τη θέση που έχει εκφραστεί στην έκθεση δραστηριοτήτων. Ουσιαστικά αναφέρεται ότι μόνο το 30% της έρευνας σέβονται τις ε, ε, προτεραιότητες που είχαν τεθεί και υπάρχει και ένας ε, μεγάλος αριθμός εμικτών φακέλων. Σε αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο των πολιτικών προτεραιοτήτων έρευνας υπήρξε μία άμεση επαφή με το Γενικό Διευθυντή που ασκείται καθήκοντα τη στιγμή και με τους επιχειρησιακούς διευθυντές και μάλιστα με, την, ε, με το τμήμα ε, της έρευνας, επιλογή και αναθεώρησης για να μπορέσουμε να διευκρινίσουμε πώς εφαρμόζονται οι προτεραιότητες που θεσπίζονται κάθε χρόνο. Η Επιτροπή ε, εντοπίζει ότι σε ό,τι αφορά το άνοιγμα των ερευνών φαίνεται να υπάρχει μια επικάλυψη από την πλευρά της Όλαφ ε, την έννοια της πολιτικής έρευνας με καθαρά νομικές απαιτήσεις όπως ε, παραδείγματος χάρη επαρκείς ε, υποψίες ή υποψίες ή της αναλογικότητας. Η πρόταση της Επιτροπής είναι να κάνει μια πολύ σοβαρή συζήτηση με το νέο Γενικό Διευθυντή της Όλαφ ε, προκειμένου να αποσαφινιστούν αυτές οι έννοιες γιατί θεωρούμε ότι δημιουργούνται εμπόδια στον ορισμό και στην εκτέλεση ε, των ε, προτεραιτήτων της πολιτικής έρευνας, ε, έχοντας κατά νου τους στόχους της δημοσιονομικής πολιτικής και τη δημιουργία της ΕΠΟ. Και λαμβάνοντας υπόψη το σημείο αυτό, και βάσει της ε, εμπειρίας της ε, Επιτροπής ε, και της πολυπλοκότητας των υποθέσεων θεωρούμε ότι θα έχουμε καλύτερα και πιο ρεαλιστικά αποτελέσματα αν ο καθορισμός των προτεραιοτήτων της πολιτικής έρευνας γίνεται, γίνει πολιετές, πολιετής. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν θα θέλαμε να καταρτιστούν οι πολιτικές τουλάχιστον σε ένα επίπεδο δύο ετών. Και θα ήθελα να πω ότι θέλουμε να επικεντρωθούμε στην ε, πτυχή της ταχύτητας των ε, ερευνών και θα είναι μια πτυχή που θα συνεχίσουμε να συζητάμε φυσικά και ε, υπό το φως του να πετύχουμε θετικά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ. With your permission, Chairman. Με την άδειά σας, κύρια Πρόεδρε, που ο να δώσω το λόγο στην άλλη συνεργάτηδα μου. Κυρία Στρονικόφσκα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε να αναπτύξουμε ορισμένα θέματα. Λίγα λόγια για την διάρκεια των ερευνών Όλαφ, που μπορεί να ενδιαφέρει την Επιτροπή σας. Η παρακολούθηση της διάρκειας των ερευνών εντάσσεται, ε, είναι μάλλον ένα από τα καθήκοντα της Επιτροπής Εποπτείας, σύμφωνα με τον κανονισμό Όλαφ. Οι έρευνες θα πρέπει να γίνονται με συνέχεια και η διάρκεια τους θα πρέπει να είναι αναλογική με τις συνθήκες της υποθέσεως, το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι καθαρά στατιστική έννοια. Είναι σημαντική διότι η, η διάρκεια της έρευνας επηρεάζει θεμελιώδη δικαιώματα των προσώπων ε, και βέβαια μπορεί να θέσει σε κίνδυνο και τη συνέχεια που δίνεται στην έρευνα από τις εθνικές αρχές και άλλα όργανα. Δεν υπάρχει σύστημα που να μπορεί να απαιτήσει κανείς την επίσημη συνέχιση μιας έρευνας του όλα από τη στιγμή που θα έχει αρχίσει. Γι' αυτό είναι υποχρέωση του Γενικού Διευθυντού να κοινοποιεί στην Επιτροπή Εποπτείας μετά την πάροδο δεκαμήνου και μετά ένα εξάμηνο την ε, πορεία των υποθέσεων. Δυστυχώς μετά από ανάλυση 470 εκθέσεων για υποθέσεις για το 2017, η Επιτροπή Εποπτείας συμβεραίνει ότι για τις περισσότερες από αυτές δεν είναι ικανοποιητική η εξέλιξη και πρέπει να διερευνηθούν οι λόγοι για την μη ολοκλήρωση των ερευνών, καθώς επίσης και για την επιτάχυνσή τους. Η Επιτροπή Εποπτείας στην έκθεσή της ζητεί από τον Όλαφ να βελτιώσει το σύστημα αναφορών του 12 μήνου και προτείνει σε συνεργασία με τον Όλαφ ένα νέο πρότυπο για την ε, κοινοποίηση των προφοριών αυτών με στόχο να επιτύχουμε συμφωνία με τον Όλαφ για το πρότυπο ε, κοινοποίηση αναφορών που να βασίζεται στο νομικό πλαίσιο λειτουργία του Όλαφ και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από την Επιτροπή Εποπτείας και από τον Γενικό Διευθυντή του Όλαφ για τον έλεγχο της διάρκειας των ερευνών. Ελπίζομαι ότι η πρόοδος για την υπόθεση αυτή θα, γίνει, θα υπάρξει σύντομα σε συνεργασία με τον νέο Γενικό Διευθυντή. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία ε, Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Μουνιός, που είναι και ο τελευταίος που θα μιλήσει από ε, εμάς. Ευχαριστώ πολύ. Είναι τιμή μου να μπορέσω να συμμετάσχω σε αυτή τη συζήτηση Επιτροπής Ελέγχου του προπολογισμού ακριβώ όπως και η συγγήτρια που είχε ασχοληθεί δύο μήνες ε, ε, είχε καινούργιο γενικό διευθυντή και εγώ το ίδιο γιατί από τον ε, Δεκέμβριο μόλις ε, εργάζομαι στην Επιτροπή φέτος και μόλις ένα μήνα το 17 εγώ είμαι αρμόδιος για τους πόρους της ε, Όλαφ, τον προϋπολογισμό της. Και ήδη έγινε μια σύντομη μνήμα αυτά τα οποία αναφέρουμε στην έρευνα όσον αφορά τα δεδομένα ο CM αυτό το κόστος της ε, διαχείρισης των ερευνών OCM τα αγγλικά λέγαμε και οπότε θα πρέπει να δούμε ακριβώς τι επιπτώσεις έχουν οι υπηρεσίες του συστήματος πληροφορικής που είναι κάτι το βασικό για την έρευνα. Και όπως προελέχθη, από αυτές τις υπηρεσίες δεν είναι 100% ικανοποιημένοι οι χρήστες. Άλλο θέμα για να ληφθεί υπόψη είναι το ζήτημα του προσωπικού. Έχουμε πρόβλημα της διάρκειας της επιλογής. Υπάρχει μια κυκλική εναλλαγή που παρά είναι ε, συχνή. Άρα θα πρέπει με κάποιο μηχανισμό να μένει περισσότερο το προσωπικό. Είναι πιο σημαντικό για μας παρά για άλλες υπηρεσίες, γιατί χρειαζόμαστε καλούς ερευνητές, ειδικού με συγκεκριμένη κατάρτιση. Ακριβώ αυτά που είπαν σήμερα το πρωί ε, κάποιοι ομιλητές. Όλο ένα και πιο σημαντικό είναι να υπάρχει τεχνική εξειδίκευση. Βεβαίω είμαστε σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και χρειάζεται το προσωπικό της Όλαφ ακριβώς λόγω των σχέσεων με την εισαγγελία να έχει πολύ ειδικέ γνώσεις. Οπότε για να μπορέσει να μείνει εξάρτητη η Όλαφ χρειάζεται επαρκής πόρος για να μπορεί να κάνει τις έρευνες για καταπολέμηση παρανομίας και απάτης. Έτσι θα ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη προς το Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα. Θα αναβαπτιστεί η αξιοπιστία της Ένωσης και θα έχουμε πιο σημαντικά αποτελέσματα σε επίπεδο οικονομικό. Θα πιάσουν τρόπο τα, τα έξοδα για την υπηρεσία μας περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. Δεν θέλω να πω ότι θα πρέπει να δώσουμε στην Ολαφχώς να ζητούμε. Βεβαίως, όλα τα όργανα τα οποία περνούν από έλεγχο και υποπτία ακριβώς όπως το Ελληνικό Συνέδριο και εσείς και εμείς που ε, κάνουμε αυτή τη δουλειά. Βεβαίω θα πρέπει να ζητούμε πολλά από την Όλαφ. Πάντως από πλευράς δικής μας Επιτροπής Εποπτείας, τουλάχιστον από τότε που ήρθα τον ε, Δεκέμβριο, ε, διαπίστωσα ότι δεν έχει αρκετούς πόρους για τη λειτουργία της η όλες δουλεύουμε στην Εποπτική Επιτροπή, έχουμε ε, άλλε υποχρεώσει επαγγελματικέ στην πατρίδα μα. Χρειαζόμαστε εδώ όμω κάποια ειδικά καταρτισμένη υπηρεσία γραμματεία για τη δουλειά μα. Εδώ. Ευχαριστώ. Okay. Γιάν Μούλτερ, αυτές ήταν οι δικές μας ε, συμβολές στη συζήτηση. Δεν μίλησαν όλοι οι παρόντες από την Επιτροπή Εποπτείας, αλλά βεβαίως όλοι στη διάθεσή σας για να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πρώτα πολύ για την έκθεσή σας που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι σημαντική. Καθώς και οι γνωμοδοτήσεις 1 και 2 για το 2017 που είναι σημαντικές για μας. Δεν έχουμε και αντίρρηση να συντάσσετε και περισσότερες γνωμοδοτήσεις. Εσείς είστε σημαντικό ελεγκτικό όργανο και το μοναδικό για τον Όλαφ που διαθέτουμε. Έχετε λοιπόν μια ιδιαίτερη ευθύνη, την οποία ε, ασφαλώς σας ενθαρρύνω να αναλαμβάνετε, διότι ο έλεγχος βεβαίως έχει και αποτρεπτικό χαρακτήρα και ο έλεγχος οφείλει να γίνεται με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Στην έκθεσή σας συναρτάτε, ή μάλλον προσαρτάτε πολλές νομοδοτήσεις. Πότε μπορούμε να περιμένουμε τις νομοδοτήσεις αυτές ε, για το ηλεκτρονικό σύστημα για υποθέσεις οι οποίες δεν άνοιξαν. Ε, μιλείτε για 64 υποθέσεις εκεί. Η πρώτη μου ερώτηση λοιπόν είναι αυτή. Πότε θα έχουμε αυτά τα έγγραφα. Δεύτερο, όταν εξετάζει κανείς την έκθεση σε λεπτομέρεια, μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει περιορισμένη πρόοδος και για ορισμένες σημαντικές κριτικές ε, του συστήματος εποπτείας, αλλά και από εμάς βλέπουμε ότι η πρόοδος είναι περιορισμένη. Θα ήθελα λοιπόν να ερωτήσω, πώς βλέπετε και πώς θα οργανώσετε το follow-up και σε συνεργασία με τον ασκούντα ε, χρέη Γενικού Διευθυντή, αλλά και με τον νέο Γενικό Διευθυντή. Γιατί είναι υποχρέωση του Γενικού Διευθυντού να ε, ανοίξει κάποια, κάποιες υποθέσεις που δεν έχουν ανοίξει. Το ερώτημα ερευνών, ε, το πώς γίνονται οι έρευνες, όλα αυτά είναι σημαντικά και σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα των εργασιών του Όλαφ. Ε, αυτές είναι οι δικέ μου ερωτήσει, αλλά ερώτηση έχει και ο κύριος Τσεχόφσκι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ μάλλον την Επιτροπή Εποπτείας ε, η οποία ήρθε να μας δει σήμερα ε, και είναι αρμόδια για τον έλεγχο και εποπτεία του Όλαφ. Ε, τελευταία έχουμε ακούσει και από αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων σχετικά με απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και γίνονται και έρευνες και κατά υψηλά ισταμένων προσώπων. Είναι καλό που υπάρχει ο Όλαφ και που ε, δεν έχει πρόβλημα να στραφεί και κατά πρωθυπουργών εάν χρειάζεστε και να πει τα πράγματα με το όνομά τους. Εάν κάτι αποτελεί απάτη, οφείλει να αποκληθεί απάτη. Και γι' αυτό διερωτώ με εν προκειμένου ως εξής. Μιλήσατε πολύ για πράγματα τα οποία θέλετε να αλλάξετε. Έχω την εξής πρόταση. Γιατί δεν δημοσιεύετε τα αποτελέσματα των εκθέσεων του Όλαφ. Εάν θέλετε να ενισχύσετε την αξιοπιστία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, κάντε ένα βήμα παραπάνω. Εμφανιστείτε πιο διαφανείς. Κοινοποιήσετε τα αποτελέσματα των εργασιών του Όλαφ και των υποθέσεων που έχουν ε, κλείσει. Είτε είναι αρνητικά είτε είναι θετικά. Δεν θεωρείτε και εσείς ότι η αξιοπιστία του πολύ επαγγελματικού αυτού οργανισμού θα ενισχυθεί με τον τρόπο αυτό. Η πρόεδρος, δεν έχω άλλον κανένα που να ζητεί το λόγο, ο κύριος Μιλντερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε πρώτη σας σημαντική ερώτηση. Πότε θα έχετε τα αποτελέσματα και τις σχετικές εκθέσεις για τα όσα κάνουμε. Θα είμαι ειλικρινής. Έχουμε πρόβλημα με την στελέχωση της γραμματείας μας. Υπάρχει ένας αριθμός κενών θέσεων. Ψάχνουμε να βρούμε λύση. Έχουμε προβλέψει για την ώρα τον Οκτώβριο να διεξαχθεί συνάντηση του Διευθυντού του Όλαφ, του επικεφαλής του προσωπικού ε, γραφείου του Επιτρόπου, του, της δικής μας Επιτροπής Εποπτείας. Βεβαίως πρέπει ο νέος Γενικός Διευθυντής του Όλαφ να εξοικειωθεί με την εργασία, αλλά ελπίζω ότι θα μπορέσουν να πληρωθούν οι θέσεις αυτές αρχής γινωμένης από το τέλος του έτους, αρχές του επόμενου έτους. Σε ό,τι αφορά τους λόγους για τις άλλες βελτιώσεις που ζητούμε, διότι συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχουν ανάγκες βελτιώσεων, δικονομικές εγγύησεις, διάρκεια των ερευνών, ε, ποσοστό επιτυχίας των ερευνών. Εμείς θα θέλαμε να αναπτύξουμε συστήματα και διαδικασίες που να μας επιτρέπουν πολύ καλύτερη εποπτεία του, του πώς εξελίσσονται τα πράγματα αυτά και να μην περιμένουμε ε, ε τυχαίες πληροφορίες που μπορεί να έρχονται, αλλά να μπορούμε να έχουμε τις πληροφορίες και να μπορούμε και να σας κοινοποιούμε και εσά όταν χρειάζεται. Ποια μπορούν τα αποτέλεσματα. Στην επόμενη ετήσια έκθεση, το ανακοινώνουμε αυτό και στην παρούσα έκθεσή μας, ότι θα αναπτύξουμε τις σχετικές δυνατότητες. Στην επόμενη ετήσια έκθεσή μας θα σας κοινοποιήσουμε ποια είναι τα αποτελέσματα των προσπάθειων που θα έχουν ολοκληρωθεί ως τότε. Θα αναπτυχθούν λοιπόν μέσα στο, στη διάρκεια του έτους η προθεσμία που προβλέπω εγώ είναι η σύνταξη της επόμενης ετήσιας εκθέσεώς μας. Για τις παρατηρήσεις του κυρίου Τσεκόφσκι, ελπίζω ότι λέω σωστά το όνομά του, βεβαίως όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος, δηλαδή από το ποσοστό επιτυχίας. Και αυτό θα πρέπει να είναι ε, σαφές. Πολλοί έχουν πει, και εγώ δεν μπορώ να απαντήσω ναι ή όχι, ότι τα ποσοστά είναι σχετικά χαμηλά και αυτά βλάπτουν την φήμη του Όλαφ. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να βελτιωθεί. Πώς ακριβώς θα το κάνουμε δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή, αλλά είναι ένα από τα ζητήματα που συζητούμε για τα επόμενα χρόνια. Ελπίζω να επανεκλεγείτε του χρόνου και τότε θα μπορέσουμε να σας τα πούμε. Ε, αν επιτρέπετε ο κύριος Κλέμεντ να λάβει το λόγο, κύρια Πρόεδρε. Αυτό που είπε ο κ. Ντεχόφσκι. Θα μπορούσα να σας τα πω στα τσέχικα, αλλά κάτι ξέρετε, θα σας τα πω στα αγγλικά. Υπάρχουν ε, δυστυχώς πολλά εμπόδια. Και πρώτα-πρώτα έχουμε διαδοχικές έρευνες που ακολουθούν τις συστάσεις της Όλαφ. Και δυστυχώς όταν αυτά προβάλλονται στα ΜΜΕ ή τέλος πάντων δημοσιοποιούνται και στοχοποιούνται ε, το, το αντικείμενο της έρευνας, αυτό είναι αρνητικό για την έρευνα. Επίσης, ο κανισμός του GDPR θα πρέπει να αντιμετωπίσουν όλοι τα θέματα που προκύπτουν και υπάρχουν και κάποια άλλα γενικά εμπόδια για διοικητική, για οποιαδήποτε άλλη έρευνα ότι με τη διαδικασία υπάρχουν ε, ε, οικονομικές ζημίες προσνομικά ή φυσικά πρόσωπα όταν γίνεται δημοσίευση των στοιχείων αυτών των προσώπων. Επίσης είναι και θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εμπλεκομένων ή των θυμάτων. Οπότε νομίζω ότι είναι καλό θέμα προς το αν υπάρχει υποψία απάτης σημαίνει ότι κάτι γίνεται. Αλλά το αν συντρέχει περίπτωση ποινικού οδηγήματος αυτό είναι μόνο θέμα αυτό μπορεί μόνο ένα δικαστήριο να το αποφασίσει. Αλλά δεν θα πρέπει να υπάρχει δημοσιοποίηση. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Άιλετ ακόμη για να τοποθετηθεί από την σκοπιά του Όλαφ για την έκθεση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στην Επιτροπή Εποπτείας για την θαυμάσια συνεργασία μέχρι τώρα για την δυνατότητα που έχω να πάω σε κάθε συνάντησή τους να τους πω ό,τι έχω να πω, δημιουργώντας έτσι έναν επικοδομητικό διάλογο που επιτρέπει αλληλοκατανόηση. Δεν προτείνουμε, δεν προτείνουμε δημοσίευση ή ασδήποτε απάντηση στην έκθεσή τους έχουν τη δυνατότητα να επαληθεύουν τα δεδομένα χωρίς να προκαταλαμβάνονται οι γνωμοδοτήσεις τους και λαμβάνουμε υπόψη τα όσα λέει η Επιτροπή Εποπτείας. Υπάρχει ένας αριθμός τομέων όπου συνεργαζόμαστε ή προτιθέμεθα να συνεργαστούμε μόλις αυτό θα είναι δυνατόν εν ώψη των πόρων και ιδίω της πάνηθος πόρων που αντιμετωπίζουν και θα μπορέσουμε να σας ενημερώσουμε πριν από την επόμενη ε, ε, συζήτησή σας. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ το τέλος της συζητήσεως αυτής θα ήθελα να σας αποχαιρετήσω, να ευχαριστήσω για τη συνεργασία. Τα τελευταία 10-15 χρόνια είχαμε κατ' επανάληψη την ευκαιρία να συζητήσουμε και να σας δούμε και στον ρόλο σας αυτός εδώ παροιμήν. Σας εύχομαι κάθε καλή τύχη για την επόμενη περίοδο της ζωής σας και παρακαλώ παραμείνετε υγιείς. Και εγώ σας ευχαριστώ, λέει στα γερμανικά ο κύριος Άιλετ πολύ ε, ευγενέ εκ μέρου σα. Για θέματα ΙΠΠΟ και όλα, έχω να πω ότι εξή, συνεχίζει η Πρόεδρο. Δεν είναι θέμα αν κανεί είναι υπέρ τη εισαγγελία ή κατά, ή υπέρ του Όλαφ ή κατά. Χρειάζεται να οργανώσουμε μια δομή, να δημιουργήσουμε μια δομή η κατα η υπερ του ολα η κατα χρειαζεται να οργανωσουμε μια δομη να δημιουργησουμε μια δομη η οποια θα ανταποκριθεί στα καθήκοντα για τα οποία δημιουργήθηκε. Αυτό είναι το σημαντικό. Και η Επιτροπή Εποπτείας τη γνωμοδότησή, γνωμοδότησή της, την οποία αναμένουμε και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεν ενδιαφέρει τόσο να, να περιχαρακωθεί ο κάθε ένας και να προχωρήσουμε σε πόλεμο χαρακομμάτων. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο κάπως δεν μου άρεσε ε, στη σημερινή συζήτηση γιατί βλέπω δύο σειρμούς να κινούνται με ταχύτητα ο ένας ε, προς τον άλλο. Δηλαδή προβλέπω σύγκρουση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχουν αμφισβητήσεις και καυγάδες διότι και οι εντολές των διαφορετικών αυτών οργανισμών είναι διαφορετικές. Να μην φτιάξουμε και ένα τομερά περίπλοκο, ε, περίπλοκο μηχανισμό, όπως λένε. Φτάσαμε στο τέλος της ε, συνεδριάσεώς μας. Ευχαρίστω θα σας ξαναδώ στις 3 Οκτωβρίου. Ε, αποχαιρετώ και τις και τους συναδέλφους των Δυτικών Βαλκανίων. Με μεγάλη χαρά σας είδαμε εδώ κοντά μας σήμερα και πολύ ευχαρίστως θα οργανώσουμε ξανά παρόμοια συνάντηση για να ακούσουμε και εσάς. Δηλαδή, έχετε εσείς να μας πείτε. Σας ευχαριστώ. Καλή ε, τύχη, καλή επιστροφή στις πατρίδες σας. Σας παρακαλώ όλες και όλους να καταλήψετε εντάχει την αίθουσα διότι έχουμε και συνάντηση των συντονιστών.